Okay, good morning, colleagues. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπω να είναι πλήρης η αίθουσα, σχεδόν πλήρης. Και μπορούμε να συνεχίσουμε την ημέρηση διαταξή μας. Ε, το επόμενο σημείο στην ημέρηση διάταξη είναι η ψηφοφορία. και η πρώτη ψηφοφορία μας είναι η γνωμοδότησή μας για το ψήφισμα το οποίο θα συνοδεύει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015. Ο κύριος Βον έχει παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του στις 23 Ιουλίου και η προθεσμία για τις τροπολογίες ήταν μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου. 18 τροπολογίες κατατέθηκαν. Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε διανατάσεως των χειρών. Εάν υπάρχει αμφιβολία θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία και για το συνολικό, την τελική ψηφοφορία, τη συνολική ψηφοφορία φυσικά θα χρησιμοποιήσουμε ως ήθιστε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Παράγραφος 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 1 τροπολογία 3 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται παράγραφος 1 α νέα παράγραφος τροπολογία 4 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. <clears throat> Παράγραφος 1. Α νέα παράγραφος. Παρά, τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Δέλτα νέα παράγραφος. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε με ηλεκτρονικά μέσα. Ψηφίζουμε για την παράγραφο 1 Δέλτα, τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. 34 ψήφισαν 18 υπέρ 16 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Σαποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 8 στην παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. Λοιπόν, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα στις προφορίας. 16 υπέρ 19 κατά. Απερίφθη η τροπολογία. Παράγραφος 2α. Η νέα παράγραφος, τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτεται. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Ήταν η παράγραφος 3 και όχι 10, συγγνώμη. Τροπολογία 10. Παράγραφος 3, τροπολογία 11. Κύριε Βόν, έχετε το λόγο. Είχα μια προφορική τροποποίηση να κάνω εδώ. Θέλω να διαγράψω την τελευταία φράση, μια συγκεκριμένη λέξη. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε, να διαγράψουμε την τελευταία φράση στην τροπολογία και έτσι θα γίνει σαφέστερο. Ευχαριστώ. Έχουμε αυτή την προφορική τροποποίηση. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Δεχόμαστε, λέει η πρόεδρος, την προφορική τροποποίηση. Δύο έχουν αντίρρηση. Εάν ένα και μόνο μέλος αντιταχθεί σε μια προφορική τροπο, τροποποίηση, λέει η κυρία Κρέλ, τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Στην Ολομέλεια διαφορετικά. Χρειάζεται 40 βουλευτές, κάτι τέτοιο ή μια ολόκληρη πολιτική ομάδα. Ας ελέγξουμε, λέει η Πρόεδρος. Τι, λένε, τι λέει ο κανονισμός. Ε, let me, explain using the rule. Να σας εξηγήσω τι λέει ο κανονισμός. Στην Ολομέλεια χρειάζονται 40 μέλη για να εμποδίσουν μία τροπολογία, αλλά στη συνεδριάση των Επιτροπών πρέπει να είναι το ίδιο ποσοστό όπως λέει το άρθρο 169.6. Μήπω μπορείτε να μα διαβάσετε το άρθρο 169.6, λέει ο κύριο ε, Αλμπερτ. Άρθρο 168. 169. για την κατάθεση και υποστήριξη των τροπολογιών. Οι τροπολογίε θα τεθούν σε ψηφοφορία μόνο αν έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε όλε τι επίσημε γλώσσε, εκτό αν το Κοινοβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αποφασίσει ούτω αν τουλάχιστον 40 μέλη εκφράσουν την αντίθεσή του. Θα αποφύγει τη λήψη αποφάσεων που θα έθεταν βουλευτέ που χρησιμοποιούν συγκεκριμένη γλώσσα σε μία αποδεκτή μειονεκτική θέση. Όταν λιγότεροι από 100 βουλευτέ παρόντε, το Κοινοβούλιο δεν δίνει να αποφασίσει εφόσον αντιτίθεται τουλάχιστον ένα δεκάτο των παρόντων μελών. Και μετά σε πλάγια στοιχεία Προτάσει του Πρόεδρου λοιπά Θα το περάσω αυτό στην Επιτροπή. Ο αριθμός των ψήφων που απαιτούνται για τη διατύπωση αντίρρηση σε παρόμοια τροπολογία ή τροποποίηση καθορίζεται με βάση το άρθρο 209 καταναλογία που εφαρμόζεται στην Ολομέλεια με στρογγυλοποίηση ανάλογα με την περίπτωση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Τρεις ψήφοι χρειάζονται, λέει ο γραμματέας. Αν σε... Δύο, δύο στην πραγματικότητα. Παρακαλώ. Ίσως, επειδή εγώ έχω, έχω θέσει αυτή την πρόταση και ίσως μπορώ να, ξε, να εξηγήσω ότι εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν χρειάζεται τώρα να συζητήσουμε για τους αριθμούς. Έχουμε ήδη τρεις ε, βουλευτές που εξέφρασαν αντίρρηση και επομένως η προφορική τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε περάσει εδώ πολύ καιρό. Πάντα ήταν ε, ένας βουλευτής που αρκούσε για να μην γίνει δεκτή μια προφορική τροπολογία. Ίσως κάναμε λάθος στο παρελθόν, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην γίνεται κάθε φορά συζήτηση. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να τα διευκρινίσει αυτά μέχρι την επόμενη ε, συνεδρίασή μας να είναι σαφείς οι κανόνες. Τώρα δεν έχει σημασία. Ίσως όμως θα είναι κάποιο πολύ σημαντικά, σημαντικό πολιτικά θέμα και θα ήταν καλό να έχουμε ήδη τη βεβαιότητα αν ο κανόνας του ενός βουλευτή που ισχύει επί 10 χρόνια έχει αλλάξει. Και εγώ συμφωνώ μαζί σα, δεν πρέπει να καταδαπανίσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να έχουμε σαφεί κανόνε στην Επιτροπή μα και ζητώ από τη Γραμματεία να διευκρινίσει για την επόμενη συνεδρίασή μας και για την επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να έχουμε την πληροφορία για το πόσα μέλη θα πρέπει να είναι εναντίον μιας προφορικής τροποποίησης. Συνεχίζω την ψηφοφορία τώρα. Παράγραφος 3, τροπολογία 11, χωριστή ψηφοφορία εδώ, σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Πέρας. 17 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται κατά συνέπεια. Δύο αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3α καινούρια, τροπολογία 12. Κατά λέει η πρόεδρος. Εννοεί υπέρ. Συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4. 4α, νέο. Τροπολογία 14. Υπέρ. Υπέρ, συγγνώμη. Είναι νωρίς το πρωί, κάνω λάθη. Υπέρ, λοιπόν. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4α νέα. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5α, νέα παράγραφος Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5α νέα. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί ολοκ... ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία. <clears throat> Ψηφίστε τώρα. Πέρας. «35 <clears throat> υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές». Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Okay. Now we continue. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Διορθωτικό προϋπολογισμός παριθμών 3 κάθετο 2014. Έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα και τόξου κτλ. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση για το διορθωτικό προϋπολογισμό 3 του 2014 που προβλέπει αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την κατηγορία 1β. Η Επιτροπή Προπολογισμών ζήτησε την γνωμοδότησή μας ε, και έδωσε προθεσμία την 3η Οκτωβρίου το αργότερο, γι' αυτό. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεσμένο. Μόνος τρόπος να το τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ήταν να διανύμουμε μέσω της γραπτής διαδικασίας το σχέδιο θεωρητικού προβολισμού και σήμερα να ψηφίσουμε. Το χρονοδιάγραμμα αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατόν να μεταφραστούν ε, τα κείμενα, να μεταφραστεί το σχέδιο αυτό. 17 Σεπτεμβρίου λάβατε από τον κύριο Όλμπριχτ το κείμενο και μπορούσατε μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου να καταθέσετε τροπολογίες και έχουμε πράγματι λάβει δύο τον αριθμό. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις. Παραγραφός 1, τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Πρέπει να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. We have 18 uh, votes. 18 ψήφοι υπέρ, 18 κατά και δύο αποχές. Απορρίπτεται επομένως τροπολογία. Λόγω των αποχώλη πρόεδρος. Mm. Παράγραφος 3, τροπολογία 2, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ναι παρακαλώ ο κύριο Όλμπριχτ ένα πολύ σύντομο σχόλιο κύριε Πρόεδρε είναι κατεπίγουσα η διαδικασία, δεν είναι αυτό που συνηθίζεται ε, να κάνουμε στην Επιτροπή μας, αλλά υπάρχει αυτό το γενικό θέμα με τις καθυστερήσεις και πρέπει γι' αυτό να δεχθούμε το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού υπαριθμών 3 το συντομότερο δυνατό. Θέλω απλά να ενημερώσω την Επιτροπή ότι η Επιτροπή Προπολογισμών αύριο συνεδριάζει με την Επιτροπή μια ειδική συνεδρίαση και κλεισμένα των θυρών, αλλά θα υπάρξει μια ενημέρωση. Και ο στόχος είναι να μάθουμε γιατί υπάρχει αυτό, αυτή η μεγάλη καθυστέρηση που οφείλεται. Θα κάνει αυτή την παρουσίαση η Κομισιόν αύριο και μπορεί κανείς να την λάβει νομίζω σε έντυπη μορφή και είναι σημαντικό να λάβουμε αυτό το έγγραφο κι εμείς για να καταλάβουμε ότι υπάρχει καθαίρεση το ξέρουμε. Γιατί, πού οφείλεται, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Είναι σημαντικό. Και Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η Κομισιόν θα μας δώσει εγγράφος αύριο μια απάντηση, μια εξήγηση. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία αυτή. Ήταν σημαντική. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό να διευκρινιστεί για ποιο λόγο χρειάστηκε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεπίθουσα διαδικασία. Έχετε δίκιο. Και βέβαια όταν λάβουμε την σχετική ενημέρωση θα την διανύμω σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Από αύριο, έτσι, από τη συνεδρία στην αυριανή. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε. Ε, έχουμε την τελική ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης και για το σχέδιο δραστικού προπολογισμού υπερθυμών Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Yes. The vote is... Πέρας ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Η τροπολογία, λέει η πρόεδρος, γίνεται δεκτή. Και ολοκληρώσαμε τώρα τις ψηφοφορίες. Προχωρούμε με το επόμενο σημείο στη μέση διάταξη. Από το σημείο 10 θα ακούσουμε μια παρουσίαση της εξωτερικής μελέτης με θέμα το ρόλο των πόλεων στην πολιτική συνοχή 2014-2020. Μπορώ να έχω την προσοχή σας παρακαλώ. πρέπει να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε με την παρουσία της μελέτης για το ρόλο των πόλεων στην πολιτικη συνοχη συνοχής 2014-2020. Η Επιτροπή ΡΕΚΙ ανέθεσε την έκθεση αυτή, τη ζήτηση τέλο πάντων, ήδη από το 2013. Το τμήμα πολιτικής B ανέθεσε την διεξαγωγή της μελέτης σε μια ομάδα από τη Βιέννη, ΜΕΤΙΣ λέγεται. Η διευθύντρια της ε, επιχείρησης αυτής ε, θα μας παρουσιάσει σήμερα τη μελέτη, η κυρία Χέρτα Τέντλινγκ Σενχόφερ. Βασικός στόχος της μελέτης ήταν να αναλύσει τον ε, αυξημένο ρόλο των πόλεων στην πολιτική συνοχή για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 με βάση το νέο πακέτο, το νομοθετικό και με βάση την εμπειρία της προηγούμενης περίοδου προγραμματισμού. Ο αντίκτυπος, τον αυξημένο ρόλο των πόλεων, ευκαιρίε, οι κίνδυνοι, επίσης έπρεπε να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης. Η παρουσίαση της μελέτης έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί έχουμε και την ανακοίνωση της Επιτροπής του Ιουλίου για τις αστικές πολιτικές περιγράφει γενικά την κατάσταση των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε και μια δημόσια διαβούλευση για το αστικό θεματολόγιο. Μετά την παρουσίαση θα δώσω το λόγο στους βουλευτές για ερωτήσεις και τώρα παρακαλώ την κυρία Σενχόπερ που δεν τη βλέπω. Α, εκεί είστε μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Αφού ολοκληρώσατε με επιτυχία τις ψηφοφορίες, ε, μπορούμε να περάσουμε σε κάτι λιγότερο πολύπλοκο που είναι οι πολιτικές και το περιεχόμενο κάποιων πολιτικών. Και βέβαια το σημερινό θέμα είναι η πόλη. Η πόλη είναι σημαντική φορή για τη διαμόρφωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Και γιατί τονώνουν την εφηβιώσιμη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της πολιτικής συνοχής. Και αυτό που μας απασχολεί σήμερα ως ερώτημα είναι αν πραγματικά η πολιτική συνοχής πραγματεύεται παρκώς και τα αστικά ζητήματα. Αυτό ήταν το αντικείμενο της μελέτης και σήμερα θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα αυτής της μελέτης. Αν καταφέρω βέβαια να βάλω μπρο το μηχάνημα. 15 λεπτά νομίζω έχω στη διάθεσή μου, πρέπει να είμαι γρήγορη. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνοψίσω κάποια μηνύματα και να μην επισέλθω σε λεπτομέρειε ή σε μεμονωμένε μελέτε περιπτώσεων. Μπορείτε να διαβάσετε εσεί, αν θέλετε τη μελέτη. Ποιε είναι βασικά, οι βασικέ προκλήσει καταρχά ε, στα αστικά ζητήματα και στην πολιτική συνοχή, τι μπορούμε να διδαχθούμε με βάση τι εμπειρίε από το προηγούμενο ε, περίοδο προγραμματισμού 2013, ποιος είναι ο ρόλος των πόλεων στη νέα περίοδο θα δούμε εταιρικέ σχέσει, επιχειρησιακά προγράμματα, για να δούμε πώς συμμετέχουν οι πόλεις και θα ολοκληρώσουμε με συμπεράσματα και συστάσεις. Βασικές προκλήσεις για τις πόλεις, λοιπόν, πρώτο σημείο. Νομίζω, και να τα πω πολύ σύντομα, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Ζητήματα με ζήτα κεφαλαίο για τις πόλεις. Οι πόλεις έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη και την ε, ανάπτυξη βιομηχανιών που βασίζονται στη γνώση. Είναι το κέντρο της μεταποίησης ε, και εκεί πραγματικά παράγεται ανάπτυξη, τεχνολογία, επιστήμες της ζωής, δημιουργικές βιομηχανίες. Στηρίζονται κυρίως στις πόλεις αυτές, ε, αυτοί οι τομείς, αλλά και το οικολογικό αποτύπωμα, η βιωσιμότητα, επίσης συναστικά ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό. Διαχείριση της ανάπτυξης αλλά και συρρήκνωση, γιατί δεν αυξάνονται οι πόλεις, συρρυκνούνται επίσης. Έχουμε και την εξάπλωση των πόλεων με τα προάστια και γενικά επηρεάζει αυτή η ανάπτυξη των πόλεων το περιβάλλον. Και έχουμε και φύλακες κοινωνικό αποκλεισμού και πόλωση. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουν οι πόλεις. Πριν σας πω όμως ποια είναι αυτά τα προβλήματα, για να δούμε εν συντομία τι εμπειρίες αντλήσαμε στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού για την πολιτική συνοχή, που γνωρίζετε όλοι σας ότι είχε να αντιμετωπίσει τα αστικά ζητήματα εδώ και πολύ καιρό. Ξεκινήσαμε με την κοινωνική πρωτοβουλία Urban. Όχι, δεν θα σα πω λεπτομέρειε. Είναι μακρά όμως αυτή η περίοδος και είχαμε συμπεριλάβει τα θέματα συνοχής στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού σε όλες μας τις πολιτικές. θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε κάποια αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Urban. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το επίπεδο φιλοδοξίας. Βέβαια, βλέπουμε κατακαιρματισμένη συμμετοχή των πόλεων, που συμμετείχαν κυρίως σε επίπεδο προγραμμάτων, έργων. Βέβαια, αυτό είναι ένα γενικό μήνυμα. Πρέπει κανείς να δει τις λεπτομέρειες για να δει τι είδους επιχειρησιακά προγράμματα μελετήθηκαν και στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, όχι τόσο στα εθνικά, είχαν πιο μεγάλο ρόλο και συμμετοχή η πόλη. Έγινε επίση μια προσπάθεια με το πρόγραμμα Τζέσικα, ε, να έχουμε ένα νέο δηλαδή χρηματοδοτικό μέσο για την αστική ανάπτυξη. Το εφάρμοσαν αρκετά κράτη-μέλη. Μέχρι το 2012 όμως ουσιαστικά άρχισε πραγματικά να αποδίδει. Η βασική επιτυχία της, ε, με το Urban ήταν ότι πραγματικά εφαρμόστηκε μια ολοκληρωμένη αστική πολιτική από κάποια κράτη-μέλη, ιδίως από τα νέα κράτη-μέλη. Και αυτό έδωσε προσθέμενη αξία. Οι νέες χώρες πήραν την παρακαμπτήριο, θα έλεγα, σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν βιώσει 15 χώρες και εφάρμοσαν πιο γρήγορα το πρόγραμμα. Τώρα θα δούμε αν η επιτυχία βασίστηκε στην ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση ή όχι. Είχαμε μια ευφυή ανάπτυξη με εστίαση τεχνολογία, είχαμε βιώσιμη ανάπτυξη. Αλλά επαναλαμβάνω, για τα χρηματοδοτικά μέσα άργησαν τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν. Ποια είναι τα προβλήματα. Ιδίω για να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική συνοχή τη πόλη. Πρώτον, τι θα πει πόλη. Δεν υπάρχει ε, έννοια ε, για το τι είναι πόλη. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους, πάνω από 500.000 κατοίκους η πόλη, πάνω από 50.000 κατοίκους. Γιατί αυτό εξαρτάται από το εθνικό πλαίσιο. Σε κάποια 50.000 ε, πόλεις με 5.000 κατοίκους είναι μεγάλες. Αλλά σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, το Παρίσι είναι μια μεγαλούπολη με εκατομμύρια κατοίκους. Υπάρχει ένα ζήτημα μεγέθους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πώς ορίζεται η πόλη. Δεύτερον, πολιτική συνοχής εστιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό στους εντόπιους φορείς, στους εδαφικούς φορείς. Οι πόλεις δεν είναι συνήθως. Υπάρχουν διοικητικά όρια. η ενδοχώρα διαφορετική από την πόλη, χωρίζεται. Διασπά κάπως τους οικισμούς. Οι πόλεις, πρώτον, δεν έχουν μετροπολιτική διακυβέρνηση και δεύτερον, δεν συμμετέχουν οι πόλεις ως αστικοί φορείς. Αυτό είναι ένα. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να αναλύσει κανείς το ρόλο των πόλεων δεν είναι μετρήσιμο εύκολο, εύκολα. Άρα πρέπει κάλλιστα να μετρήσει τις δαπάνες για να δει κανείς με την πολιτική συνοχή ποιες ήταν οι επενδύσεις που προωθήθηκαν στις μεταφορές και συγκοινωνίες, σε καθαρές μεταφορές, ολοκληρωμένα έργα. Ξέρουμε ότι το 5% των επενδύσεων πήγαν σε αστικά ζητήματα και ξέρουμε ότι 33% των επενδύσεων Πήγε στην εδαφική κατηγορία της πόλης, λέει ο Μιλήτρια. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος των πολλών στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Έχουμε έναν βελτιωμένο ρόλο και στόχευση στα αστικά ζητήματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε το δίκτυο αστικής ανάπτυξης. Στο στρατηγικό επίπεδο, στρα, ε, επίπεδο κρατών μελών, εκεί που υποτίθεται ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι πόλεις για την ανάπτυξη των συμφώνων εταιρικής σχέσης, για τη διατύπωση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και συμπληρωματική συμμετοχή στο ΕΚΤ. Είχαμε επίσης ε, δέσμευση του 5% για ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις, αστικές επενδύσεις, και είχαμε το IT και CLLD ως εργαλεία υλοποίησης. Τώρα, τι βλέπουμε. Into what's been happening until... Τι σημαίνει μέχρι τώρα με τη Συμφωνία Συντερική Σχέση για την Ανάπτυξη Πολιτικών, για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα. Αστικό θεματολόγιο. Βλέπουμε ότι δεν είναι ο ίδιος ο χειρισμός σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Ε, αυτό ήταν ένα πόρισμα της μελέτης. Η Επιτροπή προσπάθησε να αναβαθμίσει περισσότερο το ρόλο των πόλων από ό,τι φαίνεται στην περίοδο προγραμματισμού. Επηρεάστηκαν όμως τα πράγματα από τον τριμερή διάλογο. Υπήρχαν κάποιες χώρες που είχαν προοδευτική προσέγγιση σε σχέση με τα αστικά όχι όλες όμως. Υπάρχει δισταγμός, ε, επιφυλακτικότητα για τη νέα περίοδο προγραμματικού. Το 5% βέβαια έχει εκπληρωθεί. Αν θέλει κανείς ε, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, πρέπει να κάνει παραδείγματο χάρη σε μια ώρα μια απόσταση, αλλά μετά σου λέει κάποιο πρέπει αυτή την απόσταση να την κάνει σε, σε τρία τέταρτα. Πώ βελτιώνεται μάλλον σε μισή ώρα έκανε την απόσταση και εδώ πρέπει να την κάνει σε τρία τέταρτα. Άρα δεν βελτιώνεσαι. Πώ βελτιώνεσαι έτσι τη φυσική σου κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει εδώ. Μειώθηκαν ε, τα κονδύλια σε κάποια κράτη-μέλη. 5% και μπάστα. Άρα δεν βελτιώθηκε έτσι η κατάσταση. Και με επιφυλακτικότητα χρησιμοποιήθηκαν οι ευκαιρίες από τα κράτη-μέλη. Υπήρχαν κάποιοι αστικοί φορείς που ήθελαν να ασχοληθούν με τα νέα θέματα της ε, πολιτικής συνοχής, ITI, 25% ήθελαν κάποιοι δέσμευση κοντιλίων, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να εκπληρώσουν αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας. Σε κάποιες χώρες συμμετείχαν στην, περίοδο, στην διαδικασία προγραμματισμού και στα επιχειρησιακά προγράμματα οι πόλεις όπως στην Ισπανία και σε κάποιες άλλες χώρες. Εν γένει όμως βλέπουμε ότι οι πόλεις και τα αστικά κέντρα έχουν ένα πολύ μικρό ρόλο, αν έχουν κάποιο ρόλο. Τι βλέπω στα επιχειρησιακά προγράμματα. Αν εντάσσονται σε μια ευρύτερη περιφέρεια οι πόλεις, όπως την Αγγλία με το Λίτς για παράδειγμα. Δεν λαμβάνονται τόσο υπόψη δικές τους ανησυχίες. Γιατί δεν έρχονται τόσο σε ανταγωνισμό, αν θέλετε, με τις αγροτικές περιοχές, σαν ένα περιφερειακό πρόγραμμα. Καλύπτει μια πόλη, ε, όπως ε, το Βερολίνο με το Βραδεμβούργο, για παράδειγμα. Εκεί δεν λαμβάνεται υποψηφισμός. Το Βραδεμβούργο, η ενδοχώρα του Βερολίνου, δεν είναι πλέον περιοχή σύγκλησης, αλλά μετάβασης. Οπότε τα κονδύλια πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένα ε, σημεία του Βραδεμβούργου. Με αυτό το μηχανισμό ε, κάπως παρακολύεται, παρεμποδίζεται ο ρόλος των πόλεων. Και είναι πιο αισθητό αυτό Βλέπουμε έναν άξονα μόνο προτεραιότητα να εστιάζει σε αστικά κέντρα. Άρα δεν υπάρχει πλέον αστική εδαφική προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι τα βάζουμε όλα σε έναν άξονα προτεραιότητα. Αυτό βασίζεται στην θεματική προσέγγιση πλέον ε, της ε, πολιτική συνοχής. Επειδή υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις θεματικοί στόχοι, τα εδαφικά ζητήματα παραμερίστηκαν κάπως. Το ITI, αυτό το νέο εργαλείο, δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλέ στα κράτη-μέλη. Γιατί φοβούνταν τα κράτη-μέλη ότι θα είχαν μεγάλο διοικητικό άχθος με μικρό προϋπολογισμό και ότι ουσιαστικά οι αρμοδιότητες εκχωρούνταν στις πόλεις ή στις περιφέρειες και φοβούνταν ότι δεν θα έχουν την εμπειρία ούτε τα κονδύλια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πολιτική συνοχής και γι' αυτό ήταν φυλακτικά και διστακτικά τα κρατη Θα σα δώσω κάποια παραδείγματα όμω κρατών μελών που έδραξαν αυτέ τι νέε ευκαιρίε Πολωνία, ε, η οποία εισήγε τα ITIs σε κάποιες περιφέρειες, στο ΕΤΠΑ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, έδωσαν ένα ποσοστό των κονδυλίων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων έργων με εστίαση στις μεταφορές. Που θα πρέπει όμως τα προγράμματα αυτά να είναι ολοκληρωμένα, όχι μεμονωμένα. Η Πολωνία είναι ένα λοιπόν από τα παραδείγματα τα θετικά. Η Ιταλία είναι μια χώρα που επίσης εισήγαγε ένα πρόγραμμα που ασχολείται με τα αστικά ζητήματα εφής, πόλης ε, και κοινωνική καινοτομία εστίαση σε ένα νέο εθνικό πρόγραμμα. Η Βουλγαρία επίσης προώθησε τις μικρότερες κλιμακάς πόλεις. Κάποιες λοιπόν χώρες βλέπουμε ότι πλέον ασχολούνται και υιοθετούν αυτή την προσέγγιση. Η προσέγγιση των εφιών πόλεων. Τι βλέπουμε αυτή την προσέγγιση. Ότι κυρίως αφορά την ενέργεια και την κινητικότητα. Δεν καλύπτει όλους τους τομείς. Και έρχομαι στα συμπεράσματα δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν είναι λίγα τα αστικά χαρακτηριστικά της πολιτικής συνοχής και αν και έχουμε ψηλότερο μάλλον έχει μπει σε πιο μπροστινό πλάνο αν θέλετε ο ρόλο των πόλεων και πάλι ε, δεν έχει αναβαθμιστεί τόσο σε σχέση με την περίοδο 2007-2013. Και αυτός, αυτή η δέσμευση κάποιων κονδυλίων μπορεί να είναι αντιπαραγωγική σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που είχαμε χαμηλό επίπεδο δαπανών, αλλά επίσης ε, μειώθηκαν τα επίπεδα δαπανών σε άλλες περιπτώσεις. Οι νέες χώρες, τα 12 νέα προσπαθούν να εκπληρώσουν τους νέους στόχους με διάφορους τρόπους. Οι παλιότερες χώρες όμως αφήνουν εκτός της πόλης, δηλαδή είναι κολλημένες στις παλιές διαδικασίες. Συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ατζέντα για τις πόλεις και μια κοινή αστική πολιτική με συγκεκριμένα εργαλεία είναι κάτι που λείπει και είναι απαραίτητο όμως. Με την κοινοτική πρωτοβουλία είχε διαμορφωθεί αυτό το θέμα, είχε πάρει σάρκα και οστά. Αλλά η αξιολόγησή μα είναι ότι η ενσωμάτωσή του σε άλλες πολιτικές έγινε πολύ νωρί και έτσι δεν, μια, δεν αποτέλεσε μια πραγματικά νέα προσέγγιση. Συμφωνίε εταιρική σχέσης. Επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται. Ε, ε, συμφωνίες εταιρικέ σχέσει ε, υποβάλλονται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι τι γίνεται για κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη τα αστικά θέματα στην επιλογή των έργων και δείκτες ε, και κατά πόσο υπάρχουν δείκτες για την αξιολόγηση των ε, έργων. Επίσης, ο ορισμός ε, της, των προϋποθέσεων ή της αιρεσιμότητας εξάντε. Το δίκτυο ανάπτυξης των πόλεων είναι μια πλατφόρμα για τη διαμόρφωση της αστικής ατζέντας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ούτω ώστε να προωθηθεί αυτό το θέμα στην διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασχοληθούν με την εμπλοκή των ίδιων των πόλεων στην διαμόρφωση της πολιτικής. Δεν υπάρχει καμία πλατφόρμα ούτω ώστε να μπορέσουν και οι πόλεις να πούν την άποψή τους για την διαμόρφωση της πολιτικής. Ε, ολοκληρωμένες στρατηγικές δεν υπάρχουν αρκετές. Υπάρχουν κάποια προσχέδια τέτοιων στρατηγικών, αλλά Υπάρχει πολλής χώρος βελτίωσης. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε περισσότερο, να παντρέψουμε περισσότερο τις διάφορες στρατηγικές. Επίσης, πρέπει να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τις αστικές πολιτικές και να τις εντάξουμε στις πολιτικές που διαμορφώνουν διάφορες γενικές διευθύνσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι συγκεκριμένο θέμα. Μου διέφυγε το τελευταίο σημείο. Μην ξεχνάμε τους εθνικούς ε, φορείς που είναι οι βασικοί παίχτες. Σε εθνικό επίπεδο, ποιος εκπροσωπεί τα θέματα της αστικής πολιτικής. Ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς. Αυτό συνδέεται και με το αστικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα είναι ποιοι είναι εκπρόσωποι όμως των αστικών περιοχών και του αστικού δικτύου. Γιατί ασχολούνται με την εφαρμογή ε, των ε, αποφάσεων της ε, πολιτικής συνοχής και των πολιτικών για τους, τα μεγάλα αστικά κέντρα. αυτό συνδέεται με το θέμα της διαχείρισης διακυβέρνησης και την, το να δοθούν εξουσίες στις αρχές των μεγάλων αστικών κέντρων. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πόλεις και τα προάστια συχνά έχουν κοινέ αρχές. Θα πρέπει επίση να ενταχθούν τα αστικά θέματα ε, στις πολιτικές των κρατών μελών. Είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις αυτό. Σε περιφερειακό επίπεδο τώρα φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά ε, όλα αυτά εξορτώνται και από τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Θα έχει νόημα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τα δίκτυα επικοινωνίας ε, μεταξύ των διαφορών κρατών μελών και να βάλουμε την αστική ατζέντα στα έργα μέσα, να ενισχύσουμε την ανταλλαγή ε, και την συνεργασία για αστικά θέματα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, οι βασικοί παίχτες, και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν μια πραγματικά αστική ατζέντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ακούσατε την παρουσίαση, την έχετε και σε χαρτί μπροστά σας. Έχουμε ήδη ένα κατάλογο από ευρωβουλευτές που θα ήθελαν το λόγο. Ποιος θα πάρει πρώτα το λόγο, η κυρία Κρέο. Μερσή, λέει κυρία Κρέλ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκαν τόσο εντυπωσιακά αυτά τα οποία ακούσαμε. Έχουμε κάποιες προσδοκίες και νομίζω και από την πλευρά του κυρίου Επιτρόπου έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των πόλεων και όχι μόνο να συμμετέχουν οι πόλεις στην ε, διεκπαιρέωση των ε, σχεδίων αλλά και για την ε, εξιολόγηση και διεκπαιρέωση των λειτουργικών προγραμμάτων μέχρι και το κρατικό επίπεδο. Είχαμε χθε τη συζήτηση αυτή με τον Επίτροπο Χαν, ο οποίο έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο για το θέμα αυτό και έχει τονίσει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια να είναι καλύτερα ενσωματωμένες οι, οι στο σύστημα διαφθοντικών πόρων από ό,τι στο παρελθόν και είπε ότι έχουμε πρόοδο. Τώρα η μελέτη αυτή μας λέει το αντίθετο. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να θεσπίσουμε ένα συγκεκριμένο μέγεθος για τις πόλεις για να μπορούν να υπησέρχονται σε αυτούς τους μηχανισμούς. Είπαμε ότι κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια θα πρέπει να έχει την ελευθερία να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητές της και να καθορίσει ποιες πόλεις μπορούν να εμπλέκονται στα σχέδια αυτά ποιε είναι οι πόλει οι οποίε είναι σημαντικές για την ανάπτυξη κάθε περιοχής. Αυτή ήταν η θέληση που είχε εκφράσει η Επιτροπή μας. Τώρα το 5% αυτό είναι μια καινούρια είδηση το γεγονός ότι θα έχουμε λιγότερη χρηματοδότηση από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό με προβληματίζει. Γιατί εμείς είχαμε την ε, μέρημνα να έχουμε ένα πρόσθετο ποσό, να ξεπερνάμε το κατώτερο επίπεδο και θα ήθελα πραγματικά να καταλάβω σε ποιο βαθμό συναρμόζεται η μελέτη αυτή με αυτά τα οποία μας δήλωσε ο κύριος ε, Επίτροπος χθες. Ίσως θα μπορούσε να μας διευκρινίσει καλύτερα η παρουσιάστρια. Κύριε Βάισοφ, ευχαριστώ κύριε <clears throat> Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μου τα πήρε από το στόμα η κυρία Γκρέλ και με τον κύριο Άλμπρεχτ είχαμε και άλλα παραδείγματα όπου υπήρξε πρόβλημα στην πολιτική των πόλεων, υπήρξε μια αντίφαση με αυτό το οποίο είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχε καταφέρει να επιτύχει και αυτόν τα οποία άκουσα τώρα. Οι πόλεις πράγματι έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το γνωρίζουμε αυτό και είπαμε ότι μαζί με τον κύριο Επίτροπο Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία γιατί ο κύριος Επίτροπος μας είχε βοηθήσει πάντα στις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πόλεων. Φυσικά και οι περιφέρειες πρέπει, όπου ανήκουν οι πόλεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά θελήσαμε για τις πόλεις να υπάρξει μια αναβάθμιση της αντιμετώπισης τους, να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είχαν μέχρι τώρα και από το 2014 πράγματι οι πόλεις αποκτούν νέες δυνατότητε χρηματοδότηση. Εγώ έρχομαι από μια περιοχή που είναι πλούσια μέσα στα ευρωπαϊκά στάνταρ, την ε, Βαβαρία. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα μπορέσουν οι πόλεις να μπορούν να πέσουν κάποιο ρόλο στην εφαρμογή των προγραμμάτων. Μου λένε πάρα πολύ οι πόλεις της Βαβαρίας, αλλά και οι γερμανικές πόλεις. ότι είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό το οποίο προβλέπεται η αρχή της εταιρική σχέσης για τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Γι' αυτό εμείς είχαμε τονίσει ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι επιτόπιοι παίκτες μέσα σε εισαγωγικά θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα εξασφαλίσουν ότι τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου θα μπορούν να φτάνουν στον τελικό δικαιούχο που είναι ο πολίτης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για τις κοινότητες και τους Δήμους και αυτό που είπε ο κύριος Χάν είναι σωστό. Όταν μιλάμε για πολιτική των πόλεων να ξέρουμε ακριβώς τι εννοούμε. Δεν θέλουμε να έχουμε μια αντιπαράθεση πόλεων και υπαίθρου. Υπάρχει μια συνεργασία και μπορούν πράγματι να εποφεληθούν οι μεν από τους δε σε αυτή την περίπτωση. Βλέπω λοιπόν σε αυτά τα οποία είπατε μια κάποια αντίφαση έναντι αυτών τα οποία εμεί έχουμε επεξεργαστεί τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Ίσως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για όλα αυτά. κύριο Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την προηγούμενη ομιλήτρια είχα την ε, ευκαιρία να διαπραγματευτώ κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια παρεξήγηση είτε οι εθνικές κυβερνήσεις δεν διαβάζουν τους κανονισμούς ή η Κομισιόν δεν κατάφερε να εξηγήσει τι ήθελε να επιτύχει. Εμείς αυτό που θέλαμε και μάλιστα και αυτό που ήθελε το Κοινοβούλιο να κάνει η Κομισιόν. Και μάλιστα δεν αναφέρεται πουθενά και το Κοινοβούλιο. Μισέ από τι ερωτήσει που αναφέρατε δεν προέρχονται από την Κομισιόν, κυρία μου, αλλά από το Κοινοβούλιο. Επομένω, μην ξεχνάτε ότι εμεί δεν είμαστε απλοί παρατηρητέ. Ε, πολεμούμε για την αστική ατζέντα. Ε, και μερικές φορές είμαστε και πιο έμφερμοι μαχητές από την Κομισιόν. Τώρα κάποια πράγματα. Το mainstreaming ήταν λάθος. Ε, έγινε πολύ νωρίς η ενσωμάτωση της αστικής διάστασης στις διάφορες πολιτικές. Έπειτα, ε, είναι πολύ ωραία η... η τομής, είναι οι τομείς που προωθεί η Κομισιόν, οι έξυπνε πόλεις και η Γενική Διεύθυνση Regio ε, δεν συμμετείχε στην ανάλυση για τις έξυπνε πόλεις. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ε, η Εύσος πολύ είναι καλή ιστορία όμως. Υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Εσείς ε, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο, ε, το επίπεδο συμμετοχής των πόλεων είναι το ίδιο. Αλλά έτσι σχεδιάστηκε. Δεν θέλαμε να μειώσουμε το ρόλο των πόλεων. Θέλαμε να αλλάξουμε την ποιότητα της συμμετοχής. Και στο τέλος της συνδιαλλαγής, τι προτάθηκε να βάλουμε κάποια κονδύλια κατά μέρο για πιλωτικά προγράμματα. Το 5% δεν είναι, δεν είναι χρηματοδότηση για τι πόλει. Θυμάμαι κάποιο υπουργό από τη Δανία, νομίζω, κάτι να συνάντηση. Μια συνάντηση που είχε με οργανώσει, ε, είπε Ευχαριστούμε για το 5%. Εάν είναι 5% για τι πόλει, θα καταφέρουμε και χωρί. Δηλαδή, πριν είχαμε 50, τώρα έχουμε 5. Εάν είναι έτσι, είναι καταστροφικό. Το 5% δεν ήταν λεφτά για πόλεις, ήταν λεφτά για πιλωτικά προγράμματα και έτσι είναι ακόμα. Και δεν αποκλείεται να έχουμε 50, 60, 70% ας πούμε χρηματοδότηση για την πόλη, εάν το δεχτεί η περιφέρεια ή το κράτος. Το 5% τι ιδιαιτερότητα έχει. Ήταν καταρχάς συνεργασία μεταξύ πόλεων και των προαστίων. Ε, Δεύτερο στοιχείο. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και μάλιστα εγώ πρότεινα τον ορισμό ε, της πόλης που να ορίζεται με βάση τη λειτουργία τους. Δηλαδή ε, πρέπει να έχω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά πρέπει να λάβω υπόψη και τη ιδιαιτερότητα της πόλης. Τρίτο στοιχείο. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων. Υποχρεωτικά. Στο τέλος της διαλλαγής ε, είχαμε φτάσει σε μια ελάχιστη κλίμακα για την επιλογή των έργων ε, είχαμε ένα μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης και το ελάχιστο ε, το δίνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ανεξάρτητη επιλογή ε, έργων από τις αστικές αρχές. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία δηλαδή, επιλογή. Θα πρέπει οι αστικέ αρχέ να αποφασίζουν, θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότηση και θα είναι υποχρεωτικά. Τρίτον, κάτι που χρησιμοποιούμε στην Πολωνία το ITI. Δεν υπάρχουν ITI στον πληθυντικό. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 5% αλλά και στο 100%. το ITI είναι η νέα μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα προγράμματα τα οποία αφορούν πολλούς τομείς. Ε, είναι τόσο περίπλοκο που ούτε η Κομισιόν δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, το ITI. Τώρα, το ITI στο 5% μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι το ITI. Αυτή είναι η τελευταία εκδοχή του κανονισμού. Επομένως το 5% δεν βασίζεται κατά ανάγκη, δεν χρησιμοποιείται με βάση τα ITI. Στην Πολωνία εμείς αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ITI στο 5%. Αλλά το ITI είναι κάτι πολύ πιο ευρύ. Είναι ένα εργαλείο, είναι μια μέθοδος για όλη την περίοδο. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Το θέμα είναι πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτά τα πιλωτικά προγράμματα για να ενισχύσουν κάτι καινούριο, που είναι η συνεργασία, εταιρικέ σχέσει, διασυνοριακή συνεργασία και χώρες αρμοδιοτήτων. Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίσουν τα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι, μπορεί να το ρυθμίσει η Κομισιόν και να πει, κοιτάξτε, είναι στον κανονισμό, άρα πρέπει να το εφαρμόσετε. Αν ξεπεράσετε το 5%, Α, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε να δώσετε στις πόλεις, όχι ένα ελάχιστο επίπεδο, αλλά μεγαλύτερη ανεξαρτησία, μ, γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα. Η έκθεση σας δείχνει ότι ο καθένας τελικά κάνει τι θέλει. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα. Έχει τον πρώην ε, πρόεδρο τη ε, Επιτροπή των Περιφερειών και ξέρετε ποια ήταν η διαμαρτυρία τη Επιτροπή των Περιφερειών για την πλατφόρμα. Ήταν ότι πολλαπλασιάζονται τα προγράμματα. Ε, και άλλοι φορεί θέλανε, ήταν κατά αυτής της πλατφόρμας. Γιατί η Κομισιόν θέλει αυτή την πλατφόρμα. Γι' αυτό τελικά μετά από όλη αυτή την κατακραυγή που έφαγε η Κομισιόν, τη μετονόμασε ε, σε πλατφόρμα. Συγγνώμη, σε δίκτυο, σε δίκτυο. Την πλατφόρμα μετονόμασε σε δίκτυο αλλά όμως το δίκτυο ισχύει και αυτό ήταν προϋπόθεση της Επιτροπής των Περιφερειών που είπε αν θέλετε να δημιουργήσετε ε, δίκτυο θα συμφωνήσουμε ποτέ. Αν θέλετε όμως ανταλλαγή εμπειριών, οκ. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξε η Κομισιόν το δίκτυο, γι' αυτό. Αυτά και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Το βασικό ήταν να υπάρξει κάτι καινούριο. Το 5% είναι ένα, μια ευκαιρία, ε, είναι κάτι το πιλωτικό. Το ITI είναι στη διάθεση ή όχι των κρατών μελών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι, αλλά η ελάχιστη εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι υποχρεωτική. Πριν από 7 χρόνια προσπαθήσαμε στο Κοινοβούλιο να την επιβάλλουμε και απορρίφθηκε ε, από την Κομισιόν λόγω της επικουρικότητας. Τώρα τα καταφέραμε. Η έκθεσή σας δείχνει ποια είναι η κατάσταση δεν νομίζω ότι διαβάσατε και το τελευταίο κομμάτι της διαφάνειάς σας, το να, το να μην μειώσουμε ε, το smart ε, στην ενέργεια μόνο και στις μεταφορές, σωστό. Το θέμα είναι να πούμε ότι ε, εμείς, το Κοινοβούλιο, θέλουμε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν για να λειτουργήσει αυτή η σχέση. Και επιπλέον ε, υπάρχει και ο κανονισμό. Δεν μπορείτε να τον ερμηνεύετε όπω θέλετε. Θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει το 5% για τα πιλωτικά. Τα υπόλοιπα 40-50% α είναι όσο θέλει, δεν έχει σημασία. Αλλά αν κάποιο λέει ότι το 5% είναι για τι πόλει και δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τι πόλει, μόνο 5% χρηματοδότηση, δεν έχει καταλάβει καλά τον κανονισμό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρίνκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την παρουσιάστρια για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά από αυτή την παρουσίαση έχω την εντύπωση ότι η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι τόσο λαμπερή όσο θα έπρεπε να είναι. Κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα όταν ακούγα την παρουσίαση είναι το ότι Εάν η πόλη είναι τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, έχουν λιγότερη φροντίδα κατά, κάποιο, κατά αυτόν τον τρόπο. Έχω, έρχομαι από μια τέτοια πόλη. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, αν η μελέτη διεκ, διεκρύβωσε ότι είναι έτσι τα πράγματα, ποιες είναι οι συστάσεις της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τροποποιηθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι όταν μια μεγάλη πόλη βρίσκεται σε μια ευρύτερη περιφέρεια, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενσωμάτωσης και είτε είναι στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας είτε σε κάποια άλλη περιφέρεια της Ευρώπης θα πρέπει να μπορούν αυτές οι πόλεις να επωφεληθούν απόλυτα από, την αστική, από το αστικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κυρία Μάλετιτς. Σας ευχαριστώ και εγώ σύμφωνα απόλυτα με όλους τους συναδέλφους και ιδίως με τον Ιαν Άλμπερτ, γιατί νομίζω ότι έχουμε πραγματικά ένα πρόβλημα με την εφαρμογή του κανονισμού. Ζητάμε συνέχεια από την Κομισιόν να μας εξηγήσει πώς εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η εταιρική σχέση στην πράξη. Η απάντησή τους είναι το εξασφαλίζουμε γιατί το λέει ο κανονισμός και παίρνουμε και από τις εθνικές ε, κυβερνήσεις τους εκπροσώπους που μας εξηγούν με ομάδες εργασίας, πώς έχουν σε επαφή με τα διάφορα τμήματα της κοινωνίας και πώς έχουν ε, ακούσει τις απόψεις τους για να προετοιμάσουν στρατηγικού χαρακτήρα έγγραφα. <clears throat> Δεν φτάνει αυτό όμως. Πρέπει να προετοιμάσουμε εθνικά έγγραφα στρατηγικής πρώτα, που να βασίζεται όχι μόνο στην αρχή εκ των άνω προς τα κάτω, αλλά και εκ των κάτω προς τα άνω. Χρειαζόμαστε να συμμετέχουν λοιπόν οι πόλεις, χρειάζεται να εμπλέκονται και οι περιφέρειες αλλά και οι δήμοι και οι κοινότητες. Έτσι μόνο θα μπορούμε να προετοιμάσουμε στρατηγικού χαρακτήρα έγγραφα στο επίπεδο των περιφερειών και μετά στην, ε, στο εθνικό επίπεδο να συνδυάσουμε τα διάφορα επίπεδα. Σε πολλές χώρες νομίζω ότι αυτό δεν έχει γίνει και γι' αυτό καταλήγουμε τώρα με την ανάλυση αυτή όπου λέτε ότι δεν υπάρχουν ακόμα στην πολιτική συνοχή στοιχεία που να είναι ιδιαίτερα για τις πόλεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και επίσης εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ολοκληρωμένες στρατηγικές και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πράγματι είναι απαραίτητο στον κανονισμό αυτό και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί η Κομισιόν δεν επέμεινε για τις αρχές της εταιρική σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ κύριο Σίμων. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κάτι και μένα με εξέπληξε στην ε, έρευνα αυτή γιατί τα τελευταία 15 χρόνια έχω μια επαγγελματική δραστηριότητα η οποία μου δείχνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που μου λέτε και μιλάω φυσικά για τη Γερμανία από όπου προέρχεται. Υπάρχουν οι διαμαρτυρίες των Δήμων ότι δεν τους λαμβάνουν υπόψη στα λειτουργικά προγράμματα. Υπήρξαν προσπάθειες, αλλά δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα αυτή η συμμετοχή. Τώρα όμως με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Έρχομαι από τη Βάδη Βιρτεμβέργη και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι την τελευταία στιγμή μπόρεσαν και αυτοί να μπουν μέσα. Λοιπόν, δεν συμφωνώ με αυτά που είπατε ως εκπρόσωπος από την ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Και όπως είπε και μία από τις ε, ε, προηγούμενες ομιλήτριες, είπε ότι δεν υπάρχει δυσκολία να ενσωματωθούν οι πόλεις στις περιφέρειες. Έχουμε περιοχές οι οποίες έχουν κάποιες ε, δυσκολίες σε επίπεδο δομών βέβαια. <clears throat> Αλλά δεν βλέπω γιατί υπάρχει πρόβλημα να μπορέσει να ενσωματωθεί μια πόλη στην ε, περιφερειακή πολιτική μιας ευμαρούς περιφέρειας. Εγώ έρχομαι από την περιοχή του Νέκαρ και ξέρω ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν που χρησιμοποιούν και την ε, περιφέρεια, την ενδοχώρα μιας πόλης και εξακολουθούν να δίδουν και στις πόλεις ε, αυτό το οποίο χρειάζεται. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ αυτού που γνωρίζω εγώ και αυτό που λέτε εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εσείς είπατε κάτι που το παρουσιάσετε και στις ε, διαφάνειες. Είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πόλεων στην ε, ανάπτυξη πολιτικής για τα Ταμεία Συνοχής, για το, τη νέα στρατηγική του Ταμείου Συνοχής. Είπατε το Κοινοβούλιο δεν έκανε αυτό επαρκώς. Μα το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν το κάναν αυτό. Ξέρετε τι είναι η διαπαραταξιακή ομάδα Urban. Σας λέει κάτι. Δεν το ξέρετε. Έρχεστε εδώ μας παρουσιάσετε μια μελέτη όπου δεν έχετε λάβει υπόψη ένα σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής πολιτικής. Κοιτάξτε πριν από πέντε χρόνια τι είχε γίνει. Ο κύριος Όλμπρεχτ το τόνισε ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε καταφέρει να έχουμε επαφές με μικρούς και μεγάλους φορείς από πόλεις. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μια καλύτερη εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής. Πολλές λοιπόν από τις προτάσεις που ήρθαν από τη διαπαραταξιακή ομάδα Urban πέρασαν ως τροπολογίας, πέρασαν ως στοιχεία που έχει δεχτεί η Κομισιόν. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα και εσείς δεν λέτε τίποτα για όλα αυτά. Έχετε μια μελέτη που λέτε αντίθετα και αυτό εγώ το βρίσκω πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Ζέλερ έχει το λόγο. Κύριε Ζήμο, πρέπει να πω κάτι αντίθετο με αυτά που είπατε. Ακούσαμε χθες τις προθέσεις, σήμερα ακούμε την πραγματικότητα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα αν έρχεται κανείς από μια περιοχή στη Γερμανία που έχουν προωθηθεί αυτά τα πράγματα ή όχι η παραταξιακή ομάδα αυτή, η, Ουλ, η Urban που ήσασταν και εσείς και ο κύριος Σόλμπραφ ήθελε πράγματι να επιτύχει αυτά. Αλλά εγώ έχω ακούσει και από μικρές και μεγαλύτερες πόλεις στη Γερμανία ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη τους, δεν συμπεριελήφθηκαν στη διαδικασία. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η Κομισιόν όσο και τα ομοσπονδιακά κράτη της Γερμανίας θεωρούν ότι, οι μικρές πόλεις δεν έχουν την ικανότητα, την ίδια ικανότητα όπως οι μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο για να παίξουν ε, κάποιο ρόλο στην πολιτική αυτή. Διαβάστε λοιπόν τις ανακοινώσεις τύπου της Ένωσης των ε, Πόλεων και Κοινοτήτων της Γερμανίας που τονίζει αυτό το γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν μπορώ παρά να ε, επικροτήσω αυτά που λέει η μελέτη γιατί θέτει αυτό το πρόβλημα επιτάπητος. <clears throat> Αποφασίσαμε το Δεκέμβριο μια σειρά από κανονισμούς. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εταιρικέ ε, ε, συμφωνίες στη Γερμανία, αλλά αυτά βασιστήκανε στο σχέδιο της Κομισιόν και μόνο στο αρχικό σχέδιο της Κομισιόν και όχι μονάχα και όχι επί τη βάση αυτών που αποφασίσαμε εδώ. Το 2012 εγώ είχα έρθει σε επαφή με, πολλές, ε, σε πολλά ομόσποδα κρατήδια της Γερμανίας όπου συζητήθηκε το θέμα των λειτουργικών αυτών προγραμμάτων και αυτά τα είχαμε προετοιμάσει μέσα στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο είναι υπερπτουσία τώρα της ε, μελέτης είναι το γεγονός ότι καταδεικνύει ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν μπορεί κανείς να αλλάξει. Εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε πει όχι εκεί ως ε, συνομοθέτες και τελικά δεν περάσαμε την ε, θέση μας γιατί το 5% όπως είπε ο Γιάνν χρησιμοποιείται μονάχα σαν ένα άλοθη για τα μικρά προγράμματα και για να καλύψει τις ε, μικρές πόλεις και υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση της πολιτικής συνοχής. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λάβουμε ιδιαίτερα στα σοβαρά και θα πρέπει να επιμείνουμε. Η μελέτη αυτή είναι μια μελέτη που είναι ορθή σε σχέση με τις μικρές και μεσαίες πόλεις στη Γερμανία κατά την άποψή μου. Μπορεί να μην ισχύει αυτό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχουν πολλές λοιπόν πόλεις οι οποίες ε, δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να φέρουν σε πέρα στα σχέδια επενδύσεων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει δυσκολία να ενσωματωθούν σε μια καλύτερη πολιτική συνοχή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρέσο. Προσπαθήσω να θα μιλήσω ιταλικά για, για να είμαι πιο σαφής. Το θέμα των ε, αστικών πολιτικών στο εσωτερικό της περιφερειακής πολιτικής, γιατί γι' αυτό ουσιαστικά μιλάμε, αυτό είναι το σημαντικό. Παρότι υπάρχουν εμπειρίες που ξεφεύγουν από το περιφερειακό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτό λοιπόν το θέμα των αστικών θεμάτων πρέπει να το διαχειριστούμε με πολύ προσοχή. Γιατί η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια περιφερειοποιημένη πολιτική. Όχι μόνο οι στατιστικές αλλά και τα προγράμματα βασίζονται στην περιφέρεια. Η μονάδα είναι η περιφέρεια. Στην περιφερειακή είναι περιφερειακή πολιτική λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουν οι περιφέρειες. Φυσικά έχουν ε, τα κράτη ε, τα εθνικά προγράμματα, αλλά τα πραγματικά επιχειρησιακά προγράμματα είναι περιφερειακά. Έτσι. Εκτός και αν τα κράτη είναι πάρα πολύ μικρά, που διατηρούν ας πούμε, το επιχειρησιακό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο. Τα επιχειρησιακά προγράμματα λοιπόν είναι περιφερειακά και πρέπει να είναι έτσι μέσω των εταιρικών σχέσεων που έχουν ε, συνάψει με τις αστικές ε, περιοχές. Αστικές περιοχές σε κάθε χώρα είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Γιατί όλες μας οι επικράτειες ε, είναι διάσπαρτες από πόλεις. Το θέμα είναι τι εννοεί ο καθένας με τον όρο αστική περιοχή. Αν μιλάμε για μεγάλα αστικά κέντρα, είναι προφανώς ότι οι πόλεις είναι πάντα οι βασικοί εταίροι των περιφερειακών πολιτικών. Εάν τώρα κάποιος πάει να δει που, είναι, ε, που εστιάζονται οι παρεμβάσεις, σε πάρα πολλές περιπτώσεις εστιάζονται και στις πόλεις. Και επομένως, στη φάση του προγραμματισμού είναι σημαντικό η εταιρική σχέση σε περιφερειακό επίπεδο να εμπλέκει 100% με στρατηγικό τρόπο τις πόλεις. ακόμα και αν έχουν διαφορετικές διαστάσεις, γιατί έχουμε τις μεγάλες πόλεις που, που είναι σημαντικά αστικά κέντρα και φυσικών θα έχουν διαφορετικά έργα από τις άλλες πόλεις που είναι στρατηγικές, σημαντικές για την ίδια περιφέρεια, αλλά που έχουν τελείως διαφορετικές άλλε διαστάσεις. Σε τι πρέπει να χρησιμεύσει αυτό που υπενθύμησε ο Γιάνν ο οποίος υπενθύμησε τις ανησυχίες που είχε η Επιτροπή των Περιφερειών, που όπως είναι γνωστό εκπροσωπεί και τις πόλεις. Ε, ποιες, είναι, οι ανησυχίες λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών για αυτή την πλατφόρμα της ε, Κομισιόν. Φοβόταν ότι θα δημιουργήσει αντιθέσεις, ότι θα δημιουργήσει προβλήματα δηλαδή σε επίπεδο προγραμματισμού η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας. Η ανησυχία η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και με την ε, ανησυχία ότι οι πόλεις τελικά θα περιοριστούν στο 5%. Έτσι. Το οποίο δεν είναι καν λογικό, δεν είναι καν δυνατό. Τώρα, αυτό το 5% τι να πούμε γι' αυτό. Να υπενθυμίσουμε ότι αποτελεί ουσιαστικά ένα ταμείο για πειραματικά προγράμματα, για να επεξεργαστούμε νέα εργαλεία για τις αστικές πολιτικές. Και πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί πραγματικά έτσι αυτό το 5%. και να καταλάβουμε αν κάτι έλειψε στο παρελθόν και από ό,τι λέει και η μελέτη αυτή, λείψαν πράγματα ε, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα προγραμματισμού. Εδώ δεν μιλάμε για ταμεία, αλλά μιλάμε για τη δυνατότητα να πείσουμε μια νέα δυνατότητα προγραμματισμού. Και αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν είναι να μας εγγυηθεί ότι στην ε, εκπόνηση και συνεχεία την εφαρμογή των ε, περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι πόλεις εμπλέκονται 100% ήδη από τη φάση του προγραμματισμού. Και προφανώς και στη φάση χρήση των πόρων έχουν λόγο. Εννοείται. Ο πειραματισμός είναι κάτι άλλο. Και από την άλλη έχουμε την, την χρονική στιγμή ε, πραγματικής χορήγησης των πόρων, που φυσικά δεν μπορεί να περιορίζεται στο 5%, έτσι χρηματοδότηση 5% για τις μεγάλες πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι γελίο. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε από την Κομισιόν και να υπενθυμίσουμε. Να τις υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι για να είναι συνεπής συνολικά η πολιτική θα πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο, να παίξει το ρόλο της η περιφέρεια. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει ένα μικρό κομματάκι, ένα ψίχουλο. Θα πρέπει συνολικά υπεύθυνα είναι η περιφέρεια και να εμπλακούν οι μεγάλες πόλεις και κυρίως βεβαίως η πρωτεύουσα της περιφέρειας κτλ. Ήδη από την αρχή, του, από την αρχή της διαδικασίας, τον προγραμματισμό μέχρι τη χρήση των πόρων, μέχρι το τέλος δηλαδή. Ευχαριστώ ως μέλος της Επιτροπής να πάρω και εγώ το λόγο. Όχι on the, on the urban agenda. για την αστική ατζέντα. Και φυσικά θα μιλήσω βουλγάρικα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις πληροφορίες που μας ε, δώσατε με τη μελέτη. Τώρα που αρχίσαμε την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού και τώρα που διαπραγματευόμαστε για αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι πολύ σημαντική αυτή η μελέτη. Δυστυχώ, από την εμπειρία που έχουμε από το 2010-2013 για να προετοιμάσουμε την ενεργό συμμετοχή των πόλεων και την παρουσία τους στην, στον προγραμματισμό, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αρκετά απεσιόδοξοι από τη συμμετοχή των πόλεων. Στη Βουλγαρία κάναμε μια απόπειρα. Γιατί έχουμε, δημιουργήσαμε ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα για την αστική ανάπτυξη. Για το σχεδιασμό των δικτύων μεταφορών, για εκπαιδευτική υποδομή, για κάθε υποδομή στις πόλεις και για τη μετακίνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις αστικές περιοχές. Έχουμε αυτά τα πλάνα. Απλώς είναι συμπλήρωμα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης που σύναψε η Βουλγαρία. Και ο μόνος τρόπος που μπορούν να εφαρμοστούν στο μέλλον είναι να αποτελέσουν τμήμα του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο είναι υποδιαπραγμάτευση τη στιγμή που μιλάμε. Το πρόγραμμα αυτό το αναφέρθηκαν σε αυτό διάφοροι συνάδελφοι. Ο ευρύς ορισμός της πόλης ως ε, μια μεγάλη περιοχή που ορίζεται από τον αριθμό των κατοίκων είναι ένας πολύ χοντρικός ορισμός και δεν καλύπτει την αστική κατάσταση σε πάρα πολλές ε, περιοχές της Ευρώπης που διαφέρει. Όπου μπορεί να έχουμε ας πούμε πόλεις μεσαίου μεγέθους και όμως είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της περιφέρειας, επειδή είναι εκεί που είναι, Μερικέ φορέ είναι βασικό μοχλό τη ε, περιφερειακή ανάπτυξη αυτέ οι πόλει και γι' αυτό είναι σημαντικέ. Από την εμπειρία μα, ε, έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με του ορισμού για πράγματα που είναι διαφορετικά. Πόλεις, που μπορεί να είναι πραγματικά μοχλή ανάπτυξη Και με την ε, ολοκληρωμένη προσέγγιση, ε, όπου λαμβάνουμε υπόψη μας το πυρήνα της πόλης και τα προάστια, ας πούμε, τις γύρω-γύρω περιοχές που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται για την ανάπτυξή τους από τον πυρήνα της πόλης. Έχουμε απερίμωση κάποιων πόλεων, ε, υπάρχει το ανάποδο σε άλλες περιοχές, Κάποιες από τα προάστια χάνουν τις ε, λειτουργίες τους, ειδικά όταν είναι πολύ κοντά στις, ε, στα κέντρα των πόλεων. Ελπίζω ότι όταν η πολιτική αστικής ανάπτυξης εφαρμοστεί, εμείς ως Επιτροπή θα είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε την όλη διαδικασία. Χαίρομαι που χθε συμφωνήσαμε να ζητήσουμε μία μελέτη για την αστική ανάπτυξη. Μία μελέτη η οποία θα παρακολουθεί τα, τη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης και το πώς ε, εξελίσσονται τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτά τα θέματα θα τα έχουμε συνέχεια υπόψη μας και σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας ακόμα μια φορά. Έχουμε κάποιον άλλο ομιλητή. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, με, έφερε πολύ αυτή η συζήτηση και άκουσα πολλά και για το πώς όλοι εργαζόμαστε με συναντικό τρόπο. Ήταν κάπως ε, έντονες ε, ορισμένες ε, παρεμβάσεις σήμερα, με εξέπληξε αυτό. Το θέμα δεν είναι όμως να βασιστούμε στον αγγελιοφόρο, αλλά στις ειδήσει που μας φέρνει. Θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο το αγγλικό και ιδίω στα Midlands ε, και στη Βόρεια Αγγλία, στη δική μου περιφέρεια και αλλού οι πόλεις δεν λειτουργούν ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτών των ε, μέτρων, των πακέτων ε, μεταχρηματοδότηση, με ενδιαφέρει γιατί σίγουρα δεν είναι η μοχλή ανάπτυξη πάντα σε διάφορα εθνικά κράτη. Ακούσαμε και από την πρόεδρο την περίπτωση της Βουλγαρίας για την απερίμωση και στη Γαλλικία και στη Σικελία το βλέπουμε και σε άλλες περιφέρειες. Στην Αγγλία οι αγροτικές ε, πραστικές περιοχές όμως αντιθέτως είναι μοχλός ανάπτυξη, άρα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να μου πείτε αν η μελέτη εφαρμογή των πολιτικών λαμβάνει υπόψη αυτή τη σημαντική διάκριση μεταξύ ορισμένων πόλων που είναι μοχλή ανάπτυξη και κάποιων άλλων που χρειάζονται, θέλουν χρηματοδότηση βοήθεια γιατί εκεί είναι χαμηλή επιχειρηματικότητα και το επίπεδο ανάπτυξη σε σχέση με την ε, ενδοχώρα. Και επίσης ε, τα σχόλια της μελέτης για την εκπροσώπηση και τα όρια ήταν ενδιαφέροντα αυτά τα σχόλια γιατί είναι λίγο αντιφατικό το ότι και είναι και αναπόφευκτο ότι χρειάζονται φωνήμενοι πόλεις αλλά έπειτα οι ίδιοι λένε, και το καταλαβαίνω, ότι η χώρα χρειάζεται, όλοι χρειάζονται φωνή δηλαδή. Αλλά πώς μπορεί να, έχει ή να έχουν την ίδια φωνή και να ακούγονται εξίσου οι πόλεις και η ενδοχώρα. Ποιος εκπροσωπεί ποιον είναι λίγο πολύπλοκο και συγκεχημένο, αλλά νομίζω ότι αυτή η εκχώρηση αρμοδιοτήτων, ε, ιδίω στην Αγγλία, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματο στη Σκωτία για τη χώρα με τον Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένα θέμα τώρα που μα απασχολεί πάρα πολύ. Ε, ξέρω ότι έχουμε ω ομάδα δυσκολίε και κάποιε άλλε πολιτικέ ομάδε φαντάζομαι είχαν δυσκολίε. Με αυτή την έννοια και τα σχόλια που άκουσα, ότι η ρύθμιση είναι ρύθμιση και ότι πρέπει να είναι αυτό υποχρεωτικό. Μα ανησυχεί αυτό, διότι Νομίζω ότι ο μόνο τρόπο με τον οποίο μπορεί κανείς να πετύχει την αποτελεσματική εκπροσώπηση είναι να καταλάβει το εθνικό κράτος ότι είναι σημαντική η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι είναι πολύτιμη. Και αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς και πόσο μάλλον το πιο πάνω επίπεδο. Αυτέ οι συστάσει, λοιπόν για το τμήμα πολιτική. νομίζω ότι πρέπει να τα λάβει υπόψη και η Επιτροπή μας όμως επίσης πρέπει να λάβει υπόψη στο μέλλον τη διάκριση μεταξύ του μοντέλου της πόλης ως μοχλό ανάπτυξης, που ίσως το βλέπουμε στην περισσότερη, στη μεγαλύτερη Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι η πόλη ο μοχλός της ανάπτυξης. Και εκεί αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ε, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν ε, υπάρχουν ερωτήσεις, μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία Σενχόφερ για να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις ή να σχολιάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι που η μελέτη αυτή οδήγησε σε συζήτηση. Χαίρομαι για αυτή τη συζήτηση. Ήταν λιγότερο ερωτήματα, ήταν λιγότερα ερωτήματα και περισσότερα σχόλια αυτά που μου απευθύνθηκαν και θέλω και εγώ να απαντήσω για τη μεθοδολογία. Εμείς είδαμε την άλλη πλευρά. <clears throat> είδαμε δηλαδή τα λειτουργικά προγράμματα και τις εταιρικέ σχέσεις και ζητήσαμε από αυτούς που συμμετέχουν στα προγράμματα και τις εταιρικέ σχέσεις πώς πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά. Δεν ρωτήσαμε τις πόλεις λοιπόν. Μιλήσαμε σε κάποιες από τις πόλεις, αλλά είδαμε και την άλλη πλευρά. Δεύτερον, είναι κάπου 270 τα λειτουργικά προγράμματα. Δεν είναι μια μελέτη μόνο για τη Γερμανία. Και για την περίπτωση του Κίρχεν. Εγώ ήμουν παρούσα στη συζήτηση, στη συνάντηση για την εκ των προτέρων αξιολόγηση. Και τώρα πρέπει να μιλήσω στα γερμανικά. Δεν υπήρξε κανένα θέμα για την συγχρηματοδότηση από την πλευρά των πόλεων. Οι πόλεις δεν είναι εταίροι σε επίπεδο συγχρηματοδότησης. Δεν είναι αξιόπιστες πάντα και δεν ξέρουμε αν ξέρουν καλά τους κανόνες και αν μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κονδύλια γιατί υπάρχουν μεγάλες περικοπές στους προϋπολογισμούς των Δήμων και των Κοινοτήτων. Είναι πιο διαφοροποιημένη η κατάσταση αυτή λοιπόν. Και αν υπησέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες, ήταν μια επισκόπηση αυτή που έγινε και κοιτάξαμε 8 χώρες συγκεκριμένα από τις 28. Επίσης, οι κανόνες και ο κανόνας συμπεριφοράς της, ε, των εταιρικών σχέσεων διαμορφώθηκε όταν είχαν ήδη καθοριστεί οι εταιρικέ ε, σχέσεις, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας για τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων. Δεν ισχύει αυτό, λέει η κυρία Κρέλ. Η, η έννοια της εταιρικής ε, σχέσης ήταν ήδη έτοιμη στο τέλος του 2012. Γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ξέρουν ότι μια σχέση εταιρικού χαρακτήρα θα πρέπει να έχει άλλη μορφή. Το ξέραν θα αλλάξει η μορφή αυτών των σχέσεων ένα χρόνο προτού να βγει το νομικό κείμενο επισήμως. Το ξέραν τα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και το θυμάμαι πολύ καλά. Χωρίς μικρόφωνο. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής δεν είναι το θέμα της γνώσης, αλλά περισσότερο της ε, εφαρμογής. Συνεχίσουμε λοιπόν μία ακόμα πρόταση. Το θέμα της διακυβέρνηση των μητροπολιτικών αστικών χώρων είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιληθεί σε εθνικό επίπεδο. Η πολιτική συνοχή τώρα δεν μπορεί να ζητήσει μια προσέγγιση να υπάρχει, η οποία δεν υπάρχει σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί απλώ να ενισχύσει αυτή την προσέγγιση το πώς θα μπορέσουν να εξελιχθούν τα ολοκληρωμένα σχέδια, αυτό είναι ένα από τα κύρια ερωτήματα σε σχέση με την εφαρμογή των θεμάτων που έχουν να κάνουν με το θεματολόγιο των πόλεων. <clears throat> Σας ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρος. Αν δεν υπάρξουν σχόλια από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, ναι, θέλετε να πείτε κάτι. Σας ευχαριστώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με την ε, κατεύθυνση της μελέτης αυτής, αλλά έχουμε μια μικρή ανησυχία στο ότι περιγράφει κυρίως το παρελθόν και όχι το παρόν ή το μέλλον. Είναι κάπως ε, περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί. Βασίζεται κυρίως σε περιστασιακά στοιχεία εγώ δεν βλέπω να φαίνεται από αυτά που λέτε ότι ήρθατε σε επαφή με την Κομισιόν και δεν έχετε καμία μνήα επαφών με την Κομισιόν. Γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν πολλέ αντιφάσει με αυτό το οποίο γνωρίζουμε, όπω παραδείγματο χάρη η περιγραφή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων, των ITI, το τόνισε και ο κύριος Ούλμπρεθ προηγουμένω, αλλά επίση και για την ε, ε, εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Είπατε ότι είναι περιορισμένη η προσφυγή στα ITI, ενώ είναι 22 τα κρατημέλη που τα χρησιμοποιούν. <clears throat> και έχετε κάποιες γενικές δηλώσεις ότι θα είναι η ίδια η αστική διάσταση όπως ήταν στο παρελθόν. Όχι. Είχαμε μια εξέλιξη, ίσως όχι μια επαναστατικού χαρακτήρα αλλαγή, αλλά το ότι έχουμε ένα προσδιορισμό 5% χρηματοδότησης, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο το 5% που θα δαπανηθεί για την ε, ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. Εμείς θεωρούμε ότι περίπου 10% θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για μια αηφόρο αστική ανάπτυξη και όπως είπε και ο κύριος Χόλμπριχτ δεν είναι οι μόνες επενδύσεις στις αστικές περιοχές. Πάνω από 50% του Περιφερειακού Ταμείου δαπανάται σε αστικές περιοχές. Και για το ρόλο των πόλεων στις διαβουλεύσεις και τις εταιρικές συμφωνίες και πάλι νομίζω ότι είναι κάπως περιστασιακά αυτά τα οποία αναφέρονται και αποσπασματικά και δεν ισχύουν για τις περισσότερες χώρες. Για τον ορισμό του τι είναι μια πόλη, αυτό δεν νομίζω ότι ήταν πρόβλημα. Ο κανονισμός είχε ήδη μια προσπάθεια να γίνει μια λειτουργική προσέγγιση και όχι μονάχα να βασιζόμαστε στα διοικητικά όρια. Μιλάμε λοιπόν για αστικές περιοχές και όχι μονάχα για δικήτικές περιοχές πόλεων και τονίζουμε όταν υπάρχουν συνδέσεις. Η εδαφική προσέγγιση δεν περιορίζεται όπως βλέπετε στη μελέτη στο 5% γιατί υπάρχουν πολλά λειτουργικά προγράμματα που βασίζονται στην, που εστιάζουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, εθνικά λειτουργικά προγράμματα που αφορούν αυτή την περιφερειακή ανάπτυξη και έτσι ξεπερνιέται το 5%. Υπάρχουν και άλλα τέτοια θέματα και επίσης και στις συστάσεις σας νομίζω ότι είναι πεπαλαιωμένες γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαβούλευση για, μια νέα, για ένα νέο αστικό θεματολόγιο. Προσπαθούμε να οργανωθούμε στην Κομισιόν για να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών μας. Τα κράτη-μέλη συνεργάζονται για τα θέματα αυτά του αστικού θεματολογίου υπήρξε η χάρτα της ε, λειψίας και άλλα στοιχεία διακρατικής συνεργασίας και η Κομισιόν συνεργάζεται και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις πόλεις. Επομένως, ίσως θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τις συστάσεις σας με βάση αυτό το οποίο έχει γίνει στην πραγματικότητα. Εν γέννη λοιπόν είμαστε κάπως απογοητευμένοι. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δοθεί μια λαθασμένη εικόνα της πραγματικότητας με αυτή τη μελέτη και δεν έχει υπάρξει αναγνώριση των ε, βελτιώσεων που έχουν γίνει γιατί τώρα έχουμε μια πιο ισχυρή αστική και ε, παιδαφική ε, διάσταση στην πολιτική μας. Θέλετε να απαντήσετε κυρία Σιόνχοφερ. Μα είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω γιατί κάναμε μία μελέτη που βασιζόταν σε 8 κράτη-μέλη, μιλήσαμε στους εμπλεκόμενους στα λειτουργικά προγράμματα, στις εταιρικέ σχέσεις, εκπροσώπους των πόλεων. Δεν είναι μία πανευρωπαϊκή μελέτη, αυτό είναι γεγονός. Αλλά <clears throat> καταγράφω τα σχόλια της Κομισιόν και θα σκεφτούμε περισσότερο. Δεν σας κατάλαβα, χωρίς μικρόφωνο. Εντάξει, σας ευχαριστούμε. Εντάξει, το θέμα αυτό θα παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής μας και στο μέλλον και θα παρακολουθήσουμε τα λειτουργικά προγράμματα και τις εταιρικέ ε, σχέσεις και θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και για όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο για τη συμβολή τους και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο σημείο είναι η παρουσίαση της μελέτης της Κομισιόν για την, ε, μάλλον παρουσίαση της Κομισιόν για την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Είναι μία από τις πιο πρόσφατες από τις τριετούς χαρακτήρα εκθέσεις της Κομισιόν και καλύπτει την προηγούμενη γενιά ενεργειών της πολιτικής συνοχής 2007-2013 και τα συμπεράσματά της είναι ότι η περιφερειακή πολιτική έχει ανακόψει λίγο το αποτέλεσμα δικοπής των δημοσίων επενδύσεων λόγω της οικονομικής κρίσης και έχει μειώσει σε κάποιο βαθμό τις περιφερειακές ανισότητες και προσβλέπει και στην επόμενη γενιά προγραμμάτων 2014-2020 και αναφέρει πως οι επενδύσεις θα μπορέσουν <clears throat> να φύγουν από την υποστήριξη μεγάλων προγραμμάτων υποδομών για να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά προβλήματα όπως είναι η κοινωνική συμπερίληψη, η ενεργειακή απόδοση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρουσίαση αυτού του εγγράφου θα μας δοθεί από την Κομισιόν. Έχουμε δύο εκπροσώπους της DG Regio, τον κύριο Ρούντοφ Νίσλα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης για την Πολιτική και την κυρία ε, Ρίς Ντίκστρομ που είναι επικεφαλής της Μονάδος Οικονομικής Ανάπτυξης. Ανάλυσης. Κύριε Νίσλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Θέλω να σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της τελευταίας έκθεσης συνοχής. τα βασικά στοιχεία για να σας ε, σκιαγραφίσω λίγο τι έχει η έκθεση. Έχετε και την έκθεση χαρτί. Εκεί έχετε πλούσιο υλικό που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Three uh, language versions, uh, German, English and French, but you will shortly in the coming weeks have all the uh, official languages available for this report. Όλες επίσημες γλώσσες και για τις 23 και στις 23 γλώσσες. Είχαμε το φόρουμ συνοχής, ε, από αυτό προέκυψε η έκθεση και έχουμε και τον πανδέκτη αυτής της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα το έλεγα. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο της έκθεσης, απορρέει από τη συνθήκη, η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να υποβάλει αυτή την έκθεση κάθε τρία χρόνια Σε αυτή την περίπτωση της έκτης έκθεσης αποφασίσαμε να την καθυστερήσουμε λιγάκι, ούτω ώστε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της νέας πολιτικής και να τα λάβουμε υπόψη για την ε, εκπόνηση της έκθεσης. Όπως ξέρετε, η πολιτική συνοχής ασχολείται με την οικονομική ανάπτυξη. Και πρέπει να δούμε καταρχάς τα πιο σημαντικά στοιχεία, τις πιο σημαντικές τάσεις ε, που παρουσιάζει η Ευρώπη τα πιο το πιο σημαντικό στοιχείο, η πιο σημαντική τάση τα τελευταία 6 χρόνια ήταν η οικονομική κρίση. Όταν κοιτάτε αυτό το χάρτη, αποκομίστε μια διαφορετική εικόνα από ότι αν τον είχατε κοιτάξει πριν το 2008. Πριν το 2008 θα είχατε δει ότι το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ανάπτυξη σε διαφορετικούς βαθμούς από μέτρη ανάπτυξη μέχρι καλό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά τώρα η εικόνα έχει αλλάξει άρδιν και βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλος ο Νότος, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο η Ιρλανδία και η Φιλανδία Φερρυπίν, την περίοδο 2008-2011, που είχαν μια συμπίεση του ΑΕΠ. Μόνο οι πιο πλούσιες χώρες, ε, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπως Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία και κάποια από τα νέα κράτη-μέλη ε, σημείωσαν καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό οδήγησε σε κάτι που προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε μάλιστα με την πολιτική μας και ιδίως και ποιο είναι αυτό, οι οικονομικές ανισότητες, οι οικονομικές διαφορές οι οποίες ε, έχουν γίνει πιο βαθιές, πιο πλατιές από τη στιγμή που ενέσκυψε η κρίση. Κοιτάξαμε τις ομάδες χωρών όπου είχαμε την, το μεγαλύτερο τέτοιο το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αριστερά, φυσικό είναι. Οι πλούσιες ε, χώρες είχαν αναπτυχθεί με πιο αργούς ρυθμούς, ενώ ε, με την πράσινη γραμμή οι πιο φτωχές χώρες είχαν τα, τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ε, το 2009 είχαμε την πρώτη κορυφή όπου έπληξε για πρώτη φορά την Ευρώπη η κρίση και τότε βλέπουμε ότι κάποιες από τις χώρες κατάφεραν να ξεφύγουν λιγάκι από αυτό το μοντέλο συμπίεσης και να επανέλθουν σε κάποια μέτρια επίπεδα ανάπτυξης. Το καλύτερο που συνέβη είναι με τις πιο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα είμαστε ξανά στο επίπεδο του 2% ε, ρυθμού ανάπτυξης. Οι πιο πλούσιες χώρες ε, μάλιστα κατάφεραν να διαφύγουν ε, την πρώτη πτώση, την, την πρώτη άβυσο λόγω κρίσης. Αλλά ε, εκεί που είχαμε τις χώρες μεσαίου εισοδήματος, εκεί είχαμε διπλή κρίση το 2013 και μέχρι και σήμερα ε, είναι πολύ, υστερούν πάρα πολύ. Αυτές οι χώρες μεσαίου εισοδήματος, εδώ στην ε, Ευρώπη, ποιες ήταν, χώρες ήταν αυτές, οι χώρες του Νότου. Η κρίση επίσης είχε σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης της ανεργίας. Όταν κοιτάξτε, την αριστερή γραφική παράσταση, βλέπετε ότι είναι εντυπωσιακό ότι η ανεργία αυξήθηκε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εξαίρεση της Γερμανίας. Αυτή είναι η εικόνα μεταξύ του 2008 και 2012. Και οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ανεργίας, όπως ξέρετε και φαντάζεστε, είναι, ε, σημαίνει και αύξηση της φτώχειας. Η δεξιά γραφική παράσταση είναι αυτή, α, είναι η εικόνα που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια και η ανεργία θα είναι ακόμα χειρότερη τα επόμενα χρόνια. Τώρα, πρώτο συμπέρασμα. Πώς έπληξε η κρίση στα διαφορα κράτη-μέλη. Βλέπετε κάτω-κάτω στην γραφική παράσταση ότι το πρώτο κύμα το φάγαν οι νότιε χώρες της Ευρώπης και για την ανάπτυξη του ΑΕΠ καθώς και για την ανεργία. Εκείνες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης επλήγησαν χειρότερα. Μάλιστα, για την Νότια Ευρώπη ποια είναι η κατάσταση. Όλη η σύγκληση από το 1999 εξανεμίστηκε, εξαλείφθηκε από την κρίση. Έχουμε επίπεδα του ΑΕΠ που έχουν επανέλθει στα επίπεδα του 1999 και πριν το 1999 μάλιστα. Ε, μοιάζει τώρα λίγο καλύτερο το πράγμα σε τμήματα χωρών ή σε χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αργότερα, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που τα κατάφεραν να βγουν σχετικά αλόβητες από την κρίση. Όταν βλέπετε την πρώτη γραμμή, διάφορες σχετικά φτωχέ χώρες την έβγαλαν καθαρή. Τώρα, ποια είναι τα στοιχεία που προωθούν την ανάπτυξη. Η καινοτομία, η έρευνα είναι κάποια από τα στοιχεία που στάθηκα εγώ. Σε αυτό το επίπεδο η Ευρώπη υστερεί στην υλοποίηση των στόχων της επένδυσης, δηλαδή 3% στην έρευνα και τεχνολογία. Η κατάσταση είναι πολύ πιο προβληματική στα πιο φτωχά κράτη-μέλη και ιδιαίτερο στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα θα πρέπει να διδαχθούμε κάτι από αυτό. Να διδαχθούμε κάτι από το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είναι στο ύψος των φιλοδοξιών της επίσης τη διαβίου μάθηση. Έχουμε βαλτώσει. Όταν συγκρίνουμε τα στοιχεία των τελευταίων 10 χρόνων, βλέπουμε ότι ο στόχος του να έχουμε 15% όλων των υλίκων ως μετέχοντες, ως κοινωνίτης διαβίου μάθησης, διαβίου μάθησης ε, δεν πήγε καλά ε, μέχρι το 2013. Το, 2000, ε, το 2004 είχαμε, ήμασταν στο 9%, τώρα είμαστε στο 10%. Πολύ μικρή αύξηση. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση έχουμε. Επίσης, τους χάρτες πρέπει να τους δείτε με προσοχή, γιατί έχουμε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Προσοχή, προσοχή. Ειδικά, ας πούμε, ισχύει αυτό για τη Γερμανία, Φερρυπίν όπου έχουμε την επαγγελματική κατάρτιση που εξηγεί γιατί η Γερμανία ίσως δεν είναι χώρα με πράσινο χρώμα. Όταν κοιτάτε όλους τους στόχους Ευρώπη 2020 συλλήβδη, όσοι έχουν περιφερειακά στοιχεία, η καταπολέμηση της στόχιας, η εκπαίδευση, η καταπολέμηση του αποκλεισμού κτλ. Βλέπετε μια ξεκάθαρη εικόνα απασχόληση κτλ. Βλέπετε ότι υστερούμε στα περισσότερα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απέχουμε πόρο από τους στόχους. Έχουμε ε, τη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη και τις σχετικές περιφέρειες που σε μεγάλο βαθμό ε, φτάνουν σε αυτούς τους στόχους. Αλλά όλο το ανατολικό και νότιο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόρο απέχει. Κοιτάξαμε την ενίσχυση των δικτύων των μεταφορών της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διατρέξω μερικές γραφικές παραστάσεις από το 1955 μέχρι το 2030. 12, συγγνώμη. Θα ζητήσω από το συνάδελφο να τα παρουσιάσει. Α, βλέπετε εδώ ότι το χρώμα γίνεται πιο έντονο και αυτό σημαίνει ε, μεγαλύτερος, ε, μεγαλύτερη ταχύτητα ε, στο δίκτυο, στο δικό δίκτυο. Από το 55 μέχρι σήμερα έγινε τεράστια πρόοδος, αύξηση της ταχύτητας δηλαδή. Αλλά φτάσαμε σε κάποια χρονική στιγμή όπου η πολιτική συνοχής ε, ταΐστηκε με πάρα πολλά λεφτά. Ξεκινάμε τώρα ξανά από το 2001, όπου βλέπετε ότι η Βυρική Χερσόνησος ήταν σε μεσαίο επίπεδο και κάτω, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα ε, στα μεγάλα οδικά δίκτυα τότε, ενώ το 2012 βλέπετε ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα σε αυτήν την περίοδο δηλαδή. Και σε άλλα κομμάτια της περιφέρειας, ε, Νότια Ιταλία, Ιρλανδία, άλλαξαν πολλά. Αυξήθηκε η ταχύτητα δηλαδή με τον οποίο ταξιδεύουμε. Και αυτό ε, συνδέεται βέβαια με τις επενδύσεις που κάναμε χάρη στην πολιτική συνοχή. Αλλά όταν κοιτάμε τι έχει γίνει μέχρι το 2012, βλέπουμε πόσα πολλά δεν έχουν γίνει σε κάποια κομμάτια. Ειδικά στην Ανατολική και στη Βόρεια Ανατολική Ευρώπη. Όταν βλέπουμε τους στόχους για το 2030, όπου τα περισσότερα δίκτυα είναι σε κόκκινο, με κόκκινο, προφανώς δεν έχουν υλοποιηθεί, βλέπετε την τεράστια πρόκληση Άλλο τομέα όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις και εμφανίζεται με ερυθρό χρώμα. Εδώ σας έχω παρουσιάσει τα αποτελέσματα για την χρήση ανανεώσιμης ενέργειας από το περιβάλλον και, τις, ε, και τα ενεργειακά θέματα. Δείχνει το ρόλο που έχουν στη γενική κατανάλωση ενέργειας οι ανανεώσιμες ενέργειες. Και βλέπετε ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος η οποία επιτεύχθη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα, αλλά παραμένει επίσης ένα πολύ μεγάλο κενό το οποίο δεν έχει καλυφθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το στόχο του 20% και τους ειδικού επιπλέον στόχους που έχουν θεσπίσει τα διάφορα κράτη-μέλη. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα τομέα που παίζει μεγάλο ρόλο στην πολιτική συνοχή στα επόμενα χρόνια και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο τις επενδύσεις μας. Και έρχομαι τώρα Έρχομαι τώρα στο τμήμα που έχει να κάνει με το ρόλο και τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής. Τι έχουμε πετύχει λοιπόν στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, ιδίως άμα δούμε. Αν δούμε την κατάσταση λοιπόν λόγω και της κρίσης, είδαμε ότι υπήρξε μια σημαντική μείωση στα επίπεδα δημοσίων επενδύσεων. Γι' αυτό οφείλεται με σαφή τρόπο στην ε, υποχρέωση των κρατών μελών να προχωρήσουμε σε εδραίωση των δημοσιονομικών τους και λιτότητα. Αυτό το οποίο τώρα μπόρεσε να κάνει η πολιτική συνοχή είναι κάπως να παίξει το ρόλο του μαξιλαριού στη συνολική πτώση των δημοσίων δαπανών. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα χωρίς την πολιτική συνοχή η κίτρινη γραμμή δείχνει πώς θα ήταν τα πράγματα με δίχως πολιτική συνοχής και τα κονδύλια της. Τα έτη της κρίσης, τα μαύρα αυτά έτη. Και πράγματι, η πολιτική συνοχής αποτελεί τον κύριο πόρο επενδύσεων για ένα πολύ μεγάλο μέρος των ε, κρατών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αριστερό τμήμα της ε, γραφική παράσταση βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιε χώρε για τι οποίε εκπροσωπεί πάνω από 80% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τις χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης οι οποίες μπήκανε καθυστερημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου είναι φυσιολογικό αυτό το επίπεδο, βλέπετε και χώρε όπω είναι η Πορτογαλία που ξεπερνάει το 60% και η Ελλάδα και η Ισπανία επίση με πολύ ψηλά επίπεδα. πολιτική συνοχή έχει επιτύχει πολλά. Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής για την περίοδο 2007-2013, αυτά είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Αν δείτε πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, 600.000 περίπου, μας λένε πολλά. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι χάθηκαν και 3.000 θέσεις εργασίας. Λόγω της κρίσης. Μπόρεσε να βοηθήσει λοιπόν η πολιτική συνοχή, αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει πλήρω τα αποτελέσματα τη κρίση. Υπήρξε ισχυρή εστίαση στο να υποστηρίξουμε τις εταιρείε με περίπου 80.000 εταιρείε startup σε στάδιο κίνηση που χρηματοδοτήθηκαν από την πολιτική συνοχή και υπήρξε και σημαντικό ε, αντίκτυπο στι υποδομέ 270.000 χιλιόμετρα δρόμων που κατασκευάστηκαν και επίσης το Κοινωνικό Ταμείο με 50.000 συμμετέχοντες στα διάφορα συστήματα επανεκπαίδευσης και απόκτησης προσόντων. Όταν πρόκειται επίση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουμε τις εταιρείε μέσο ενός συνολικού ποσού περίπου 13 δισεκατομμυρίων. Σε αυτό το γράφημα εδώ βλέπετε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης στα κρατη δείχνει πόσο επιτυχή είναι τα κράτη-μέλη στο να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι και να τους υλοποιήσουν σε συγκεκριμένα επενδυτικά προγράμματα. Αυτά είναι στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα. Έχουμε περίπου 215 χώρες σε όλο τον κόσμο που εμφανίζονται σε αυτό το γράφημα. Και εδώ στην ε, γραμμή που είναι του μέσου όρου βλέπετε περίπου την μέση απόδοση των κυβερνήσεων σε αυτές τις χώρες. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι τουλάχιστον στο μέσο όρο και οι περισσότερες είναι πολύ καλύτερες σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από ότι οι άλλες χώρες που βρίσκονται στη στατιστική αυτή της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας. Βρισκόμαστε και στην κορυφή του γραφήματος αυτού, στο δεξιό άκρο. Οι πιο φτωχές μας χώρες όπως είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι αυτή τη στιγμή στο μέσο όρο των 215 ε, Αν δείτε τώρα όμως, πέρα από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, βλέπετε και άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο πλούσιες και παρόλα αυτά είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Ιταλία και Ελλάδα με αρνητική τάση μεταξύ του 1996 και του 2012. Δεν θέλω λοιπόν να προχωρήσω περισσότερο σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε το πώς μια χώρα μπορεί πράγματι να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τα κονδύλια που έχουν στη διαθεσή τους για να τα μετατρέψουν σε επενδύσεις. Και στο γράφημα αυτό μπορείτε να δείτε τον συσχετισμό. Από τη μία πλευρά βλέπετε τις χώρες άνω δεξιά, οι οποίες έχουν την καλύτερη βαθμολογία στην ε, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησής τους και στο κάτω ακρό βλέπετε τις χώρες οι οποίες πόρο απέχουν από κάτι τέτοιο. Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία. Γιατί η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση σε αυτό το γράφημα. Υπάρχει μια απλή εξήγηση. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε προγράμματα εξυγίανσης εδώ και πολλά χρόνια και έχει πάρει και πρόσθετες πληρωμές και υπήρξαν και πολλές προσπάθειες από την ε, ειδική μονάδα για την Ελλάδα για να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των σχεδίων. Γι' αυτό η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίπτωση θέση. Στο γράφημα τουλάχιστον. Ερχόμαστε τώρα σε ένα τμήμα το οποίο συμπεριλάβαμε όταν εξηγήσαμε προηγουμένως τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισης στην πολιτική συνοχής. Η πολιτική συνοχής δεν είναι μια πολιτική η οποία λειτουργεί εν κενό αέρος. Λειτουργεί μέσα σε μια τριγωνική σχέση με άλλες πολιτικές. Την αντιλαμβάνομαι ως την κυριότερη πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να αντανακλά περαιτέρω τα δεδομένα της δημοσιονομικής εξαγίανσης. Οφείλει να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη ακόμα και όταν οφείλουν να περιστύλουν τους προϋπολογισμούς τους. Είναι εκεί για να μπορέσει να βοηθήσει τις δαπάνες που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη, αλλά έχουμε και την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που συνδέει την οικονομική διακυβέρνηση με αυτούς τους τομείς επενδύσεων. Στα δεξιά βλέπετε τα στοιχεία της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που είναι αναπόσπαστο στοιχείο στην ε, νέα κατεύθυνσή μας και οι κανόνες μας τονίζουν ότι η δημιουργία ικανότητος, ιδίω όπως φάνηκε και από την προηγούμενη διαφάνεια, είναι ένα κέριο θέμα και οι διαρθωτικές αλλαγές όπως τις ε, εξετάζουμε παίζουν κάποιο ρόλο στην εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Όλα αυτά εξετάζονται και στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που είναι ο πυρήνας επισκοπικού χαρακτήρα όλου αυτού του τριγώνου. Βρισκόμαστε εν μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού αυτή τη στιγμή και παρά το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα λειτουργικά προγράμματα έχουν υποβληθεί από τις ε, ε, από το Κοινωνικό Ταμείο και τα, το Περιφερειακό Ταμείο έχουμε αυτή τη στιγμή 310 προγράμματα που έχουν υποβληθεί και προς το παρόν έχουμε μόνο έξι λειτουργικά προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε ό,τι αφορά την, ε, τις ε, δαπάνες για αυτά τα προγράμματα έχουμε μια καλύτερη εστίαση στη, στο τι κάνουν τα διάφορα διαφορετικά ταμεία. Οι προτεραιότητες 1 με 4 είναι αυτές όπου επενδύει περισσότερο το Περιφερειακό Ταμείο, αλλά έχουμε και τα θέματα της ε, κλιματικής αλλαγής, την ε, αποδοτικότητα της ενέργειας. Υπήρξαν μέτρα πρόληψης των κινδύνων στον τομέα του περιβάλλοντος και εδώ υπάρχει φυσικά χαμηλότερη χρηματοδότηση. Βλέπετε όμως από την άλλη πλευρά ότι το Κοινωνικό Ταμείο έχει θέσει σαφείς στόχους για τις προτεραιότητες 8 έως 11 και το Ταμείο Συνοχής στην κλασική του μορφή τονίζει περισσότερο τις υποδομές και την διασύνδεση των υποδομών. Μόλον τούτο βλέπετε ότι το, ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο είναι αυτό το οποίο παραμένει το ουσιαστικότερο εργαλείο και ακριβώς παίζει συμπληρωματικό ρόλο με αυτά τα οποία χρηματοδοτεί το κοινωνικό ταμείο όταν είναι απαραίτητο να υπάρξει η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Όπως είχαμε επίσης σχεδιάσει, και αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε από τον απολογισμό των διαπραγματεύσεων, έχουμε πετύχει μια σημαντική εστίαση στους τομείς που έπρεπε, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, να ενισχυθούν οι θεματικές προτεραιότητες. Έλαμε με τέσσερα έχουν <clears throat> ανέλθει από το 31% στο 38% και βλέπετε και οι προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό ταμείο και αυτές ενισχύονται. Υπήρξε μείωση στις, στους περιφερειακούς τομείς που έχουν να κάνουν με τις υποδομές δικτύου, κυρίως ε, αυτοκινητόδρομοι και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Εδώ υπάρχει μια σχετική μείωση δεν είναι ακριβώς έτσι αν δείτε τα απόλυτα οικονομικά ποσά τα οποία έχουν αυξηθεί. Και όταν προεκβάλλουμε τον αντίκτυπο της νέας αυτής πολιτικής στο μέλλον, <clears throat> βλέπουμε ότι <clears throat> θα υπάρξει μια σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ σε μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εκεί όπου εστιάζονται οι κύριοι πόροι της πολιτικής συνοχής. Αλλά και πάλι θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία θα μπορέσουν να προκύψουν, τα παράπλευρα θετικά αποτελέσματα λόγω της εμπορικής σχέσης που έχουν αυτές τις περιοχές, γιατί η πολιτική συνοχή δεν επενδύει μονάχα στον πλούτο των πόλεων και των περιφερειών, έχει σαν αποτέλεσμα η Ευρώπη να αναπτύσσεται ενοποιημένα περισσότερο και να υπάρχει μεγαλύτερη ε, παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που παράγει ένα δευτερογενές αποτέλεσμα συνοχής. Θα πρέπει να θυμόσαστε αυτό που σας έδειξα στο προηγούμενο slide, ότι οι υποδομές οι οποίες και τα δίκτυα υποδομών της πολιτικής συνοχής ε, θα ενισχύσουν περαιτέρω την ολοκλήρωση της αγοράς την οποία επιθυμούμε. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν για τη συνέκθεση για την πολιτική συνοχή. Δεν τελειώνει εδώ η ιστοριούλα μας. Θα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που μπορούμε να σας φέρουμε σε σχέση με αυτά που κάνουν οι πολιτικές μας. Το επόμενο βήμα είναι το τέλος του 2017 που θα έρθουμε με μια πλήρη έκθεση για την ε, διαδικασία προγραμματισμού και θα σας εξηγήσουμε τι προέκυψε από την άσκηση στην οποία αποδεθήκαμε με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα λειτουργικά προγράμματα και τις εταιρικέ σχέσεις. Θα έχουμε επίσης στο τέλος του 2015 μια πλήρη αξιολόγηση της προηγουμένης περίοδου προγραμματισμού 2007 με 2013 που θα περιλαμβάνει σε βάθος ανατομή θεματικών ζητημάτων, εδαφικών ζητημάτων και Και μετά το 2016, εάν θέλει ο Θεός, θα έχουμε μια ενδιάμεση επισκόπηση της πολιτικής μας στον τομέα της συνοχής και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση για, τις, για την ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Και φυσικά υπάρχει και η 7η έκθεση συνοχής η οποία θα εκδοθεί το 2017 και η έκθεση αυτή θα συμπεριλαμβάνει προτάσεις σε επίπεδο πολιτικής για την χρονική περίοδο μετά από το 2020. Αυτά λοιπόν. Αυτό είναι το μέλλον σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις που θα προελθούν για την πολιτική συνοχή και σας ευχαριστώ τα μάλα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την πολύ αναλυτική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, θέλετε το λόγο, ερωτήσεις έχετε ή τα ξέρουμε όλα ήδη για την έκθεση και συμφωνούμε με τις συστάσεις και τα συμπεράσματα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ερωτήσει. Σα ευχαριστούμε πολύ. Very interesting. Do we? Oh, I'm sorry. Α, έχουμε. Παρακαλώ. Η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση μονάχα. Εγώ βλέπω ακόμα να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα με την αύξηση της ένδυας και της ανεργία σε ορισμένε περιοχέ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για μένα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατά προτεραιότητα και εκεί μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο οι διαρθρωτικοί πόροι για την αντιμετώπιση αυτή τη ένδυα. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ πολύτιμα που πήραμε από την έκτη έκθεση για τη συνοχή. Κάτι το οποίο δεν αναφέρατε είναι το θέμα των δημοσίων υπηρεσιών, των βασικών υπηρεσιών που αναφέρονται και στην Ευκή Βίβλο και που τονίζουν τη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των δημοσίων υπηρεσιών ρίου χαρακτήρα που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και ένα δεύτερο στοιχείο που δεν αναφέρεται είναι η σημασία της πράσινης ε, οικονομίας και το πόσο είναι σημαντικό να παίξουν ρόλο σε τοπικό επίπεδο. Αναφερθήκατε στι τοπικέ ε, επιχειρήσει, αλλά δεν έχετε πει πάρα πολλά για τι επιχειρήσει, οι οποίε ε, αναπτύσσουν, στον τομέα τη οικονομία χαμηλή περιεκτικότητας σε άνθρακα. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι παραπάνω στον τομέα Ευχαριστώ. Ερωτήσεις άλλες. Δεν το βλέπω. Οπότε σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαστε και στην καλύτερη κατάσταση ό,τι αφορά την δεθεσιμότητα δεδομένων για τις δημοσίες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με τη Eurostat, ε, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, μήπως μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να εφοδιαστούμε με καλύτερα στοιχεία στο μέλλον. Αλλά η συγκεκριμένη δυσκολία ήταν στοιχεία σε υποεθνικό επίπεδο που δεν είχαμε, γιατί η πολιτική συνέχιση όπως γνωρίζετε είναι μια πολιτική που εξετάζει αυτή τη διάσταση κάτω από το εθνικό επίπεδο και δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλά στοιχεία για αυτό το επίπεδο μέχρι στιγμής. Thank you, thank you very... Μάλιστα, σας ευχαριστούμε θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την παρουσίαση. Συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο σημείο της που είναι μια ακόμη παρουσίαση από την Επιτροπή. Μένει μαζί μας ο κύριος Νίσλ για να μας παρουσιάσει τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή μάλλον για τις, ε, την μακροοικονομική αιρεσιμότητα με βάση τα όσα ενέκρινε τον Ιούλιο η Κομισιόν. Ένα θέμα η μακροοικονομική αιρεσιμότητα πολύ επίμαχο. Τελικά εγκρίθηκε ο, ο, το νομοθετικό πακέτο για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα 2014-2020. Η Κομισιόν βέβαια τότε είχε υποσχεθεί ότι μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ ως αυτού πακέτου θα δώσει στη δημοσιότητα κατευθυντήριες οδηγίες. σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Διαθροτικών και Επενδυτικών Ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Αργότερα όμως από τα πεσχημένα παρουσίασε και εφάρμοσε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές κομισιών. Τέλος πάντων θα σας δώσω το λόγο για να μας εξηγήσετε τι Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. you the Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που υποβάλαμε. Πρώτα απ' όλα όμως, αν μου επιτρέπετε, και επειδή γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό ήταν επίμαχο, έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε τώρα 23. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό το άρθρο. Για να το καταλάβουμε θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα άρθρα, κοντινά αυτού στον κανονισμό. Το άρθρο 23 αφορά την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων του ESI και βέβαια έπονται τα άρθρα 24 και 25, τα οποία ασχολούνται με την αύξηση των πληρωμών για τα κράτη-μέλη, με προσωρινά δημοσιονομικά ελλείμματα και με τεχνική υποστήριξη για τα κράτη που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό γιατί σας το λέω από τώρα. Σας το λέω γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί αυτό το άρθρο 23 να αποτελεί απειλή για τα κράτη-μέλη. Αλλά όπως σας ε, εξηγώ σχετίζεται και με άλλα άρθρα του κανονισμού που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη στήριξη προ τα κράτη που αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές δυσκολίε. Αν έρχομαι στο άρθρο 23, το θέμα ήταν να δούμε αν αυτά τα ταμεία, η ΕΣΑΙ, τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά και Επενδυτικά Ταμεία, είναι αποτελεσματικά. Προβλέπεται επίση ότι τα προγράμματα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν. Φυσικά και υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αν δει κανεί την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, 2014-2020 ε, και τη συγκρίνουμε με την προηγούμενη περίοδο, 7-13, θα δούμε ότι τότε, την προηγούμενη περίοδο, υπήρχαν διατάξεις ε, που συνέδεαν ε, αυτά τα ταμεία, αλλά το Ταμείο Συνοχής μόνο τότε με τη μακροοικονομική κατάσταση και με τη διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος. Το 2014-2020 έχουμε μια πλήρη ε, προσέγγιση, δηλαδή πρέπει να υπάρχει πλήρης συνέπεια και με τις συστάσεις αναχώρα που αποφάσισε το Συμβούλιο. Περιλαμβάνονται όλα τα Ευρωπαϊκά Διαφορετικά και Επενδυτικά Ταμεία και τα σχετικά μέσα και μηχανισμοί μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες, ε, υπερβολικό έλλειμμα, οικονομικά προγράμματα προσαρμογής. Όλες αυτές οι διαδικασίες λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, είναι πιο αυτόματη η διαδικασία σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτό τι σημαίνει. Μπορεί αυτά που λέγονται να οδηγήσουν σε μηχανικές αντιδράσεις για την υλοποίηση ορισμένων προσαρμογών. Επίσης ό,τι αφορά τις δυνατότητες που προβλέπονται για με συμπληρωμών πληρωμών, συγγνώμη για την αναστολή των πληρωμών και των υποχρεώσεων. Το 23 έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τον αναπρογραμματισμό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο επαναπρογραμματισμός είναι κάτι που γίνεται συχνά στο πλαίσιο της ε, υλοποίησης των διαθετικών ταμείων. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Συζητούν δηλαδή η Κομισιόν για κράτη-μέλη κάποιες προσαρμογές στα επιχειρησιακά προγράμματα. Ακόμη και αν δεν υπάρχουν ε, έκτακτες περιστάσεις. Με το άρθρο 23 λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με μια έκτακτη περίσταση. Δηλαδή όταν ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει υπόψη τη εκβάσεις των συζητήσεων την ανάγκη προσαρμογής ε, ενδεχομένω των προγραμμάτων. Τότε, τελευταία ε, λύση είναι να γίνει να ζητηθεί μάλλον από το κράτος μέλος, από, να του ζητήσει η Κομισιόν αναπρογραμματισμό. Που μπορεί όμως και το ίδιο το κράτος να πάρει την πρωτοβουλία γι' αυτό. Ανά πάσα χρονική στιγμή. Όπως επίσης μπορεί ένα κράτος μέλος να εξηγήσει ίσως ότι έχει άλλα μέσα για την αντιμετώπιση ορισμένων προγραμμάτων. Όταν ένα κράτος μέλος ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιήσει εθνικούς πόρους για να λύσει ένα πρόβλημα, νομίζω ότι τότε η Κομισιόν δεν θα έχει αντίρρηση. Αν όμως φτάσουμε σε αυτό το σημείο και χρειαστεί α, επαναπρογραμματισμός, αν υποβληθεί τέτοιο αίτημα δηλαδή από, τα, από την Κομισιόν αλλά δεν αντιδράσει θετικά το κράτος μέλος, υπάρχει και εδώ η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του άρθρου 23. Στο δεύτερο, είναι πολύ αναλυτική διατύπωση και εκεί εξηγείται πολύ συγκεκριμένα πώς τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία επηρεάζονται από αιτήματα ε, που προκύπτουν από τη διαδικασία της ε, διακυβέρνησης. Στο δεύτερο σκέλος βλέπουμε κάποιους μηχανικούς μοχλούς, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω έτσι. Και εκεί έχουμε ένα πρέπει. Ε, δεν μιλάμε πλέον για τη δυνατότητα της Κομισιόν. Η Κομισιόν κάνει το ένα το άλλο το παράλληλο. Εμείς όμως καλύπτουμε με την ανακοίνωσή μας το πρώτο σκέλος, δηλαδή συζητούμε γιατί ή πώς, ποιες είναι τέλο πάντων ε, οι μέθοδοι διατυπώσεις για την υποβολή αιτήματο περί αναπρογραμματισμού από την Κομισιόν. Δεν αναφέρομαι καθόλου στο δεύτερο σκέλος του άρθρου 23 σε αυτή την ανακοίνωση. Και αν δείτε αυτή την ε, ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2013, και το παράρτημα συγκεκριμένα, θα καταλάβετε ότι εμείς αυτό που κάναμε ήταν να υποβάλουμε μια τεχνική επεξήγηση. Πώς δηλαδή θα ρονταριστεί και θα αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο νέος μηχανισμός. Δεν υπησέρχεται η ανακοίνωση συγκεκριμένα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πολιτικό επίπεδο, το πολιτικό σκέλος. Εμείς είχαμε ως στόχο να παραμείνουμε στα τεχνικά ζητήματα. Αν δείτε λοιπόν το παράρτημα, υπάρχει ο στόχος η Κομισιόν να εξηγήσει πώς θα εφαρμόσει τις νομικές διατάξεις στην πράξη. Τι θεωρούμε δηλαδή αποτελεσματική ή μη αποτελεσματική δράση μετά την απάντηση που λάβαμε από το κράτος μέλος. Τι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή των πληρωμών. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί το επίπεδο αναστολής. Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό το οποίο ισχύει, δηλαδή οι συστάσεις αναχώρα, όλα αυτά αντιμετωπίζονται στην τωρινή διαπραγματεύση των λειτουργικών προγραμμάτων και των εταιρικών σχέσεων. Για το λόγο αυτό δεν πρόκειται να εγκρίνουμε λειτουργικά προγράμματα τα οποία παραγνωρίζουν συγκεκριμένες συστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη χώρα. Στο τέλος του χρόνου λοιπόν ή στην αρχή του επόμενου χρόνου θα έχουμε ένα σχετικά σταθερό σημείο εκκίνησης και ο αναπρογραμματισμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο μετά από αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή συγκεκριμένα από το 2015 μέχρι το 2019. Δεν μπορεί να φτάσει ως το 2020 γιατί είναι το τελευταίο έτος της περίοδου προγραμματισμού αλλά αν αντιμετωπίσουμε το ερώτημα του τι θα γίνει μετά την διαδικασία προγραμματισμού, αυτή είναι η απάντησή μου. Και στην ε, ανακοίνωσή μας, αυτό το οποίο θέλαμε να δείξουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται ιδιαίτερα στο νομικό κείμενο, αυτό που θέλαμε να δείξουμε λοιπόν είναι ότι η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ προσεκτικά τις εξουσίες της για τον επαναπρογραμματισμό έχουμε τον σαφή στόχο της προτίμησης της σταθερότητος έναντι των συχνών αλλαγών. Ξέρουμε ότι σε διοικητικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να εμπλακούμε σε μια διαδικασία όπου αλλάζουν οι στόχοι συνέχεια. Γι' αυτό έχουμε μια σαφή δέσμευση από τη μεριά της Κομισιόν ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα. Για να δώσω μια περιγραφή, μια αδρή περιγραφή των κανόνων του παιχνιδιού. Οι αιτήσει για τη χρηματοδότηση μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τα διαφορετικά ταμεία, είτε το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Αλίας και Θαλασσίων Θεμάτων, Περιφερειακό, Κοινωνικό ή Ταμείο Συνοχής. Ή επίσης μπορούν να καλύπτουν εγκάσια τα διαφορετικά ταμεία. Και φανταστείτε ότι έχετε μια χώρα η οποία έχει εκτεθεί σε σημαντικούς κλειδονισμούς που έχουν συνέπειες στην αγορά εργασίας, παραδείγματος χάρη, εκεί μπορεί να είναι απαραίτητη πρόσθετη πόρη σε επίπεδο κοινωνικού ταμείου και τότε θα πρέπει να υπάρξει μια μετακίνηση πόρων από το Περιφερειακό Ταμείο στο κοινωνικό ταμείο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένα αγκονάρια τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά. Το ελάχιστο ποσοστό στο κοινωνικό ταμείο, οι οροφές για το περιφερειακό ταμείο και οι κατηγορίες χρηματοδότησης που ισχύουν για την ε, καταβολή, για την ε, προσδιορισμό κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές κονδυλίων δεν μπορούν να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να φύγουν από τις, τα κονδύλια από τις φτωχές χώρες και να πάνε στις πλούσιες. Η διαδικασία επαναπρογραμματισμού προβλέπεται να λάβει χώρα μέσα σε ένα διάστημα 11 μηνών. Επομένως, θα λάβει χώρα μέσα σε ένα και μόνο κύκλο αναθεώρησης της πολιτικής. Θα μπορέσει να κλείσει πρωτού ξεκινήσει ο επόμενος κύκλος και ξεκινάει με την αίτηση ενδεχομένως της Κομισιόν να υπάρξει επαναπρογραμματισμός μέσα σε τέσσερις μήνες και μετά από την έγκριση από την πλευρά του Συμβουλίου των αναχώρα ειδικών συστάσεων. Η αίτηση της Κομισιόν θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη <clears throat> και αιτιολογημένη. Θα πρέπει να είναι σαφής η ανάγκη να υπάρξει μια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εξηγείται πώ η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει για να αντιμετωπιστούν οι κείμενε προκλήσει και το γιατί οι, οι τωρινέ χρηματοδοτήσει είναι ανεπαρκεί. Εναπόκειται στην Κομισιόν να δείξει και να εντοπίσει τις πολιτικές και τις τομείς που θα πρέπει να ενισχυθούν. Αλλά τα κάτι μελη είναι αρμόδια να πούν πού μπορούν να υπάρξουν περικοπές κονδυλίων. Γιατί πολλές φορές έχουμε τα δοχεία και τα κρατημέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα επομιστεί τη μείωση. Αλλά η Κομισιόν πάντα πρέπει να είναι σε θέση να πει ότι κάποιες προτεραιότητες θα πρέπει να, να προστατευτούν από οποιαδήποτε περικοπή. Μπορεί να προκύψουν καταστάσεις όπου υπάρχει η πρόθεση να μειωθεί η χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο εργαλείο και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις. Αν έχετε μια υπερθερμασμένη οικονομία, η οποία έχει μια έκρηθμη οικοδομική δραστηριότητα, ίσως μπορούμε προσωρινά να μειώσουμε τις ε, συμβολές στον τομέα αυτό και όχι να δημιουργήσουμε περαιτέρω θησαλίδες. Και αυτό λοιπόν είναι ένα θεωρητικό παράδειγμα, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μόνο ένα ελάχιστο αριθμό προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών ε, προγραμμάτων που περικόπτονται. Δεν είναι ένας έξυπνος τρόπος αυτό, σίγουρα, να ενισχύσουμε ε, μία προτεραιότητα ή ένα πρόγραμμα και πώς κόβοντας ε, την πρικοδότηση σε όλα τα άλλα προγράμματα ή τις προτεραιότητες. Είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε σαφώς αυτό από πλευρά Κομισιόν έχει δοθεί σαφής ένδειξη για το ελάχιστο περιεχόμενο των αλλαγών. Θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη ποια είναι η φύση της παρέμβασης, ο στόχος που πρέπει να υλοποιηθεί και πρέπει να, ποια πρέπει να είναι το ελάχιστο ποσοστό των χρηματικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν ή να μειωθούν κάποιες προτεραιότητες. Η απάντηση τώρα σε όλα αυτά από τα κράτη-μέλη είναι ότι θα έχουμε έναν αναθεωρημένο πίνακα οικονομικών, ε, αναθεωρημένο πίνακα των αποτελεσμάτων, μια στρατηγική των προγραμμάτων και μια εξήγηση για το πώς θα πετύχουν τις προκλήσεις, καθώς και μια περιγραφή του είδους και παραδείγματα των δράσεων. Δεν ζητάνε από τα κράτη-μέλη να κάνουν μια νέα εκ των προτέρων αξιολόγηση. Θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν θέλουμε να γίνει όλο αυτό μια γραφειοκρατική άσκηση. Τι γίνεται αν ένα κράτος μέλος δεν αντιδράει στο αίτημα της Κομισιόν. Πρώτον, πιστεύουμε ότι μια και είμαστε σε κατάσταση μόνιμου διαλόγου με τα κράτη-μέλη, κανονικά δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αν παρόλα αυτά ένα κρατος και δεν απαντάει μέσα στις προθεσμίες, τότε αυτό αποτελεί μία, μία αποτελεσματική δράση. Δεύτερον, εάν πάρουμε την απάντηση με ένα από τα κράτη-μέλη και όταν κοιτάμε την ποιότητα της απάντησης, προκύπτει σαφώς ότι δεν είναι ικανοποιητική, τότε και αυτή θα τη θεωρήσουμε μη αποτελεσματική δράση. Και εδώ μπορούμε να έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος δεν απαντάει επί του θέματος δηλαδή δεν απαντάει στην ερώτηση που του κάνουμε ή δεν είναι συνεπές στις απαντήσεις του, λέει τη μία έτσι την άλλη αλλιώ. και αυτό παίζει εις βάρος του κράτους μέλους. Είναι εις βάρος του κράτους μέλους. Πάντως τελικά πρέπει να πούμε είτε, ή δεν υπάρχει, είτε δεν υπάρχει απάντηση, είτε δεν απαντάει το κράτος στην ερώτηση που τέθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, η Κομισιόν μπορεί να προτείνει αναστολή ενός τμήματος ή όλων των πληρωμών ενός προγράμματος ε, ή των προτεραιοτήτων, ή εν λόγω δηλαδή προτεραιότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί, όπως σας είπα, όταν ένα από τις δύο περιπτώσεις ισχύουν, δηλαδή καμία δράση ή ανεπαρκής ποιότητα της απόκρισης του κρατούς μέλους. Τότε η Κομισιόν μπορεί να προτείνει την αναστολή Η, η απόφαση όμω ε, αυτή της Κομισιόν δεν θα πάρθει έτσι ελαφρά την καρδία. Θα κοιτάξουμε δηλαδή σε τι φάση είναι το κρατό μέλο και αν είναι εξαιρετικέ συνθήκες, αν η χώρα ας πούμε είναι σε ύφεση ή αν υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά εργασία. που απαιτεί που απαιτεί να μην ε, κάνουμε κι εμείς, ας πούμε, οποιαδήποτε πράξη που θα πλήξει περαιτέρω την αγορά αυτή εργασία ή το κράτος η μέλος, τότε μπορεί η Κομισιόν να κάνει τίποτα. Τώρα, για τα κριτήρια των προγραμμάτων. Κοιτάμε τα κριτήρια για να αποφασίσουμε αν τα προγράμματα θα ανασταλούν ή όχι. Προφανώς δεν θα αλλάξουμε μης ενός προγράμματος ή μιας προτεραιότητας που θέλουμε να ενισχύσουμε. Γιατί θα ήταν παράλογο κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν θα πειράξουμε προγράμματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να προασπίσουμε, να υπερασπιστούμε και να διασφαλίσουμε, εν πάση περιπτώσει, πάση θυσία. Θα ζητήσουμε απλώς να βρεθούν οι κατάλληλοι τομείς της προτεραιότητας του προγράμματος που θα περικοπούν χωρίς ε, αρνητικές επιπτώσεις το ανώτατο όριο για την αναστολή πληρωμών είναι το 50%. 50% είναι το maximum και θα υπάρχουν και κάποια ελαφρυντικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη που μπορεί να χαμηλώσουν αυτό το ποσοστό του 50%. Όμως, σε μια περίπτωση, στην περίπτωση που το κράτος μας αντιδρά καθόλου και το Συμβούλιο αποφασίζει να προβεί σε αναστολή. Ακόμα και όταν έχει ληφθεί απόφαση αναστολής και το κράτο μέλο πάλι δεν αντιδρά, τότε μπορεί να αποφασιστεί ότι η αναστολή αυτή θα αγγίξει το 100% των πληρωμών το, της προτεραιότητας ή του επιχειρησιακού προγράμματος. Τέρμα, δηλαδή, οι πληρωμές. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβετε τώρα ότι έχω μια προσέγγιση η οποία λέει ότι θα Κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε μια αποτελεσματική δράση. Και η απάντησή μας είναι αναλογική σε όλη αυτή την προσπάθεια προγραμματισμού. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα πράγματα μηχανιστικά. Θα πρέπει να αναλύουμε τα πράγματα ανά περίπτωση για να έχουμε τη σωστή απο... απόφαση. Και είναι σαφές επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή. Ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Αν έχω μια χώρα που υποφελείται μέσω μιας μεγάλης χρηματοδότησης από αυτά τα ταμεία και απο... αποφασίσουμε την αναστολή για αυτή την με τον κανόνα του 50% μπορεί να σταματήσουν οι πληρωμές για πολύ μεγάλα ποσά. Έτσι. Εδώ η Κομισιόν θα εφαρμόσει τις ασφαλιστικές κλίδες. Ότι δηλαδή θα αποφύγουμε να τιμωρήσουμε μεγάλους δικαιού, πολλούς δικαιούχους, αν, ε, πώς θα γινόταν αυτό, ε, αν αποφασίσαμε μηχανιστικά, μπορεί να τους τιμωρούσαμε. Θα το προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Επίσης, όταν λαμβάνουμε αυτές τις αποφάσεις, πάντα λαμβάνουμε υπόψη το πώς θα περιορίσουμε την επίπτωση σε την ανεργία, στους ε, φτωχούς κτλ. Όμως, όταν το κράτος μέλος κουνηθεί και πάρει ε, κάποια απόφαση, Πάρα αυτά η Κομισιόν θα άρει την απόφαση αναστολή. Δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω διαδικασία. Σημαίνει ότι οι πληρωμέ θα συνεχιστούν να ρέουν. Δηλαδή θα δοθεί πληρωμή από την Κομισιόν σε όλα τα αιτήματα πληρωμής. Δεν θα έχουμε πια το πρόβλημα που είχαμε παλιά. Αυτές οι ροές πληρωμών, δηλαδή μπορούν να συνεχίσουν αμέσως μετά μία αναστολή, μετά μία, από μία άρση αναστολής. Τώρα, έφτιαξα και αυτή τη διαφάνεια, εδώ που βλέπετε, γιατί στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σας είπα, Υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία της ερώτησης. Υπάρχει η πολιτική διάσταση και υπάρχει και η τεχνική διάσταση και προσπάθησα να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε από τεχνική σκοπιά πάντα. Είναι σαφές βέβαια ότι όλα αυτά που κάνουμε για την εφαρμογή του πρώτου τμήματος του άρθρου 23 με το στοιχείο του αναπρογραμματισμού. Τι κάνει εκεί η Κομισιόν, ενημερώνει πάρα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν η συζήτηση με ένα κρατό μέλος οδηγήσει σε μια κατάσταση που ενεργοποιείται κάποια απόφαση, παίρνετε κάποια απόφαση, δηλαδή αναστολή, και αναστολή γίνεται πότε, όταν δεν αντιδράσει το κρατός μέλος μετά από μια αίτηση της Κομισιόν για ένα προγραμματισμό ή όταν υπάρχουν άλλες δράσεις, όπως αυτέ που υπάρχουν στο δεύτερο τμήμα του 20 αν δεν υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική δράση ε, για μακροοικονομικές ανισορροπίες, ε, θέμα ε, ελλείμματος, μη συμμόρφωση στα αιτήματα του προγράμματος μακροοικονομικής αναπροσαρμογής, όταν υπάρχει διαδρομολόγηση ε, για τη διαδικασία της αναστολής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται. Η Κομισιόν ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες των ταμείων αυτών και των προγραμμάτων που μπορεί να είναι αντικείμενο αναστολή. Πληρωμών. Ούτω προκύπτει ότι οι προβλέψεις του κανονισμού θα υλοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Θα πράξουμε ότι είναι ανθρωπίνο δυνατό για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις αιτήσει σας σε σχέση με το θέμα αυτό. Ηλίου φαϊνότερον επίση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη δική του πρωτοβουλία μπορεί να ζητήσει από την Κομισιόν ένα διαρθρωμένο διάλογο για την εφαρμογή του άρθρου 23, είτε επί μεμονωμένων περιπτώσεων, είτε δε εφαρμόζουν το άρθρο 23 έως σύνολο. Προβλέπεται επίσης στον κανονισμό ότι το 2017 η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει αναφορά σε σχέση με την εφαρμογή του ομονίμου αυτού άρθρου και εάν προκύψει η ανάγκη θα προχωρήσει στην ε, τροποποίηση ορισμένων στοιχείων των κανόνων αυτών φυσικά με μια νομοθετική πρόταση. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο λεπτομεριακή σας παρουσίαση και την παρουσίαση της ανακοινώση της Κομισιόν. Ξέρω ήδη και το γνωρίζω ότι ο κύριος Όλμπριχτ θέλει να λάβει το λόγο. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Όχι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλα αυτά τα οποία είπατε, αλλά έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, κατανόησα σωστά ότι αν υπάρξει αναστολή αν υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής και έχουμε ένα κράτος μέλος το οποίο έχει προβλήματα. Ανεργία, μείωση του ΑΕΠ. Η αναστολή θα βασίζεται στην πραγματική κατάσταση, δηλαδή δεν θα είναι ένα είδος ε, κύρωσης. Αν μια χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αποδυναμωμένη, ακόμα και αν κάνει κάποια σφάλματα, θα παραμείνει δεν θα εφαρμοστεί η αναστολή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάνει λάθη μια χώρα, το πρόβλημα είναι ότι είναι ε, αποδυναμωμένη. Αυτό κάνει πολύ σχετικές τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις έχουν σημασία και αποτέλεσμα όταν είναι αντικειμενικές κυρώσεις. Όταν ε, είναι τόσο σχετικοποιημένες οι κυρώσεις μπορούμε να μιλάμε για ντεμεκ αναστολές, για ψεύδο αναστολές. Το επόμενο ερώτημά μου είναι πόσο θα χρειαστεί για να υπάρξει στη νέα δημοσιονομική περίοδο αναπρογραμματισμός. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχανισμό, είναι απαραίτητο να έχουμε μια διαδικασία ταχεία, ταχείας έγκρισης. Γιατί αλλιώς η διαδικασία αναστολής θα καθυστερήσει και τον αναπραγματισμό. Πώς θα κάνει λοιπόν ταχύτερη τη διαδικασία αυτή η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπρεσό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα το κείμενο να μου δοθεί, παρακαλώ, της ανακοίνωσης, το συντομότερο δυνατόν, για να μπορέσω να το διαβάσω, έτσι με την ησυχία μου. Μία ερώτηση, αν κατάλαβα καλά. Η αναστολή συνδέεται ή με καθυστέρηση στον αναπρογραμματισμό, έτσι, ή με το ότι δεν εφαρμόζεται ο αναπρογραμματισμός ή τρίτον ή αφού έχει γίνει ο αναπρογραμματισμός, δεν έχει γίνει σωστή ανακατανομή των πόρων. Μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, έτσι. Δηλαδή, για να τα καταλάβω καλά. Ζητάνε από το κράτος να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα, ούτω ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό. Έτσι. Εάν δεν το κάνει, σταματάνε οι πληρωμές μέχρι να προσαρμοστεί στο αίτημα. Αλλά ακόμα και όταν κάνει τον αναπρογραμματισμό το κράτος, μπορεί να γίνει πάλι αναστολή των πληρωμών, μέχρι να προβεί το κράτος στην ε, ανακατανομή των πόρων, να πάνε δηλαδή οι πόροι σε νέο πρόγραμμα ή σε άλλο κομμάτι του προγράμματος. Αυτό εγώ κατάλαβα, θέλω να μου το εξηγήσετε για να δω αν κατάλαβα καλά. Ναι, να <clears throat> προσθέσω το ότι υπήρχε μια ε, υπήρχε ένα σύνδεσμος διαδικτύου για το έγγραφο αυτό, στο βασικό έγγραφο που σας δώσαμε και ουσιαστικά η δημοσίευση του εγγράφου αυτού είναι στο τέλος Ιουλίου. Η κυρία Βάνα. Ευχαριστώ και εγώ μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση. Μπορείτε να μου καθορίσετε καλύτερα το ρόλο των εταίρων στην περίπτωση του επαναπρογραμματισμού. Πώς η σχέση εταιρικού χαρακτήρα εφαρμόζεται σε περίπτωση επαναπρογραμματισμού. Άλλες ερωτήσεις? Όχι, δεν υπάρχουν. Α, ο κύριος Ζέλεο. Δεν έχουμε μονάχα κράτη τα οποία έχουν ομόσπονδη δομή, αλλά και κράτη τα οποία είναι συγκεντρωτικού χαρακτήρα στη διοίκησή τους. Και στο παρελθόν είδαμε ήδη ότι υπήρξε λόγω οικονομικών συνθήκων επαναπρογραμματισμός και τότε οι κεντρικές κυβερνήσεις ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία οικειοποιήθηκε όλα τα κονδύλια και επομένως χρησιμοποιήθηκαν αυτά για στόχους εθνικού συμφέροντος αλλά όχι προς όφελος των περιφερειών. Μη είπατε τώρα ότι ο επαναπραγματισμός θα γίνεται σε θα πρέπει να αιτείται σε εθνικό επίπεδο λόγω των οικονομικών συνθήκων. Μα τι θα γίνει τότε με τις περιφέρειες στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και πώς θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια σε σχέση με σχέδια τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω οικονομικών δυσκολιών και δεύτερον μπορούν να υπάρχουν εθνικές επιρροές οι οποίες θα τροποποιήσουν τις προτεραιότητες, θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις προτεραιότητες για, σε περιφερειακό επίπεδο. Σας λέει παραγωγικά ένα κράτος ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε υποδομές ε, για ευρυζωνικό διαδίκτυο και συμφωνούν και κάποιες ε, περιφέρειες σε μια τέτοια ρύθμιση, αλλά αυτό τροποποιεί τις ε, προδιαγραφές κάποιου λειτουργικού προγράμματος. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, με ποιο τρόπο μπορούν να υπάρξουν αυτές οι τροποποίησεις ώστε να, υπάρχει, να μην υπάρξει πάρα πολλή χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες αυτές αλλαγές. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις. Όχι άλλες ερωτήσεις. Κύριε Νίσλερ αν μπορείτε Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο καλά. Να ξεκινήσω από τον κύριο Ολμπρίχτ. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι θα πρέπει να κάνετε μια διάκριση. Έχουμε δύο σκέλη, το ένα και το δύο. Το δύο δεν το συζητάμε σήμερα. ούτε στην παρουσίασή μου. Και απαιτούνται αυστηρές μηχανικές, αν μπορώ να τις πω έτσι, όταν μιλάμε για αναστολή πληρωμών ή αναλήψεων υποχρεώσεων. Ωστόσο, το πλαίσιο είναι διαφορετικό, δηλαδή μια χώρα δεν έχει ανταποκριθεί σε επανειλημμένα αιτήματα του της Επιτροπής για να προβεί σε προσαρμογές. Τώρα έρχομαι στους κανόνες που προβλέπονται υπό το σκέλος 1, που έχει να κάνει με τις συστάσεις αναχώρα. Το πρώτο είναι ότι στην πολιτική μας ασχολούμαστε μόνο με τις σχετικές συναφείς συστάσεις αναχώρα. Υπάρχουν πολλές δηλαδή συστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις ε, επενδυτικές προτεραιότητες που είναι δικό μας αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Πρέπει τώρα να εντοπίσουμε κατά πόσο τα επενδυτικά ταμεία είναι τα καταλληλότερα, αυτά πρέπει να κινητοποιηθούν, αλλά μπορεί το κράτος μέρος να μην συμφωνεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μπορεί τότε να ζητηθεί επαναπρογραμματισμός. Και από αυτή την πλευρά, και έτσι απαντώ νομίζω και στο ερώτημα για τις καθυστερήσεις, τι θα γίνει με τις καθυστερήσεις κτλ. Τότε ξεκινά διάλογος με το κράτος μέλος. Και το πρώτο βήμα σε αυτό το διάλογο είναι καταρχάς μια άτυπη απάντηση που περιμένουμε από το κράτος μέλος. Και μετά εμείς διατυπώνουμε ως Κομισιόν τις παρατηρήσεις μας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αν αυτή η ανταλλαγή δεν οδηγεί προ σωστή κατεύθυνση, δηλαδή είτε προ την εξέβρεση μια λύση που είναι εκτό του πλαισίου πολιτική μα. και εμεί εδώ εμένουμε στο πεδίο και στο πλαίσιο τη πολιτική μα. Ε, αλλά δεν έχουμε την κατάλληλη απάντηση. Τότε θα πρέπει πλέον επισήμω τα κράτη-μέλη να υποβάλουν απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα έχει χαθεί ένα σημαντικό βήμα. Μία φάση δηλαδή στη διάρκεια τη οποία θα μπορούσε να έχει εξευρεθεί λύση. Αν τώρα δεν έχουμε είτε καμία αντίδραση, είτε η αντίδραση που έχουμε δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, η Κομισιόν υποβάλλει αίτημα αναστολής πληρωμών. Και στην προκειμένη περίπτωση προβλέπεται ότι λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση του κράτους μελ. Αλλά οι πληρωμές τι σημαίνει. Επίσης ότι αναστέλουμε τις πληρωμές για τα σχετικά αυτά ε, σκέλη του επιχειρησιακού προγράμματος. Δηλαδή μελετούμε πού μπορούμε να αναστείλουμε πληρωμές χωρίς, πώς να το πω, να δυσκολεύσουμε ακόμη περισσότερο τα κράτη-μέλη που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολία. Άρα υπάρχει ένα είδος διαφοροποίησης και διαβάθμισης για να μην τιμωρήσουμε τα κράτη-μέλη που ζητούμε να αναλάβουν δράση. Τώρα αυτό που θέλω να είναι σαφές είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν μια θετική της Κομισιόν. Τώρα η όλη διαδικασία πόσο μπορεί να κρατήσει, το πολύ 11 μήνες. Γιατί μετά είμαστε κοντά στον κύκλο του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου και έχουμε τις νέες στάσεις αναχώρα. χώρα. Θα σας πω όμως και τι βλέπουμε την ε, μέχρι στιγμής εμπειρία μας. Οι συστάσεις αναχώρα πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει από το ένα έτος στο άλλο. Δηλαδή είναι συνήθως πολυετής. Άρα μπορώ να φανταστώ μόνο μια πολύ έκτακτη περίσταση. Για παράδειγμα, να έχουμε αντιμετωπίσουμε το εξή. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης ενέργειας στις χώρες, παραδείγματος χάρη της Ανατολής λόγω των εξέλιξεων στη γεωπολιτική κατάσταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πολύ έκτακτη, ίσως ναι πράγματι θα έπρεπε κάποιος να κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει αυτή την ε, κατάσταση. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει σύσταση. για να κοιτοποιηθεί η στήριξη προ ορισμένου τομεί ή περιοχέ. Όμω, κανονικά, υπό φυσιολογικέ συνθήκε, αυτέ οι συστάσει χώρα έχουν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωή, αν μπορώ να το πω έτσι μέχρι ό,τι εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Και έχουμε εξαντλήσει όλα τα θέματα για την κυρία Μπρέσο. Δεν ξέρω αν την κατάλαβα καλά, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που ζητεί ένα προγραμματισμό. Όμως, ενεργούμε βάσει των εντολών του Συμβουλίου. Δηλαδή χωρίς συστάσεις του Συμβουλίου δεν φτάνουμε σε αυτή τη διαδικασία όπου μπορεί η Κομισιόν να επιμείνει για έναν επαναπρογραμματισμό. Γνωρίζετε βέβαια ότι είναι σύνδεση πρακτική να γίνονται συζητήσεις για κάποιες προσαρμογές των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου που έχουμε με τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άρα έχουμε πράγματι και σαφή συσχέτιση με τις στάσεις αναχώρες Για τον, για τον Αυστριακό. Α, η κυρία Μπρέσο θέλει να διευκρίνηση. Ναι. Όμως στο τέλος μιας διαφάνειας λέτε ότι αν συμφωνήσει το κράτος στην αλλαγή αναστέλλεται η πληρωμή μέχρι να αλλάξει το κράτος μέλος την κατανομή των πόρων του. Την κατανομή των πόρων από, πρόγραμμα σε πρόγραμμα δηλαδή. Όταν λοιπόν συμφωνήσει με τον αναπρογραμματισμό η αναστολή θα μπορούσε να συνδέεται και με την αλλαγή κατανομής των πόρων. Δηλαδή, ναι, λέει το κρατός μέλος, θα αναπρογραμματίσω. Δεν έχει ανακατανείμει τους πόρους από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Παρ' αυτά θα προβείτε στην αναστολή. Αυτό εγώ κατάλαβα. Αλλά ίσως δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά, τη διάβασα ή εν δεν, κα... δεν... έτσι τα ερμήνευσα αυτά που διάβασα. Να διευκρινίσετε Ναι, ακούστε. Αν έχουμε μια κατάσταση που σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε χρήματα από ένα πρόγραμμα μεταφορών, για παράδειγμα, όπου εκεί είναι μεγάλα συνήθως τα κονδύλια, για να κάνεις κάτι στον τομέα, ας πούμε, της εκπαίδευσης. Αν είναι σαφές, αυτό που λέω, δεν αναστέλουμε τα κονδύλια για το πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό. Α, ναι, το καταλάβατε. Εντάξει, λοιπόν, τα κράτη-μέλη αν συμφωνήσουμε αυτή την αλλαγή, έχουμε άρση του αδιεξόδου και της αναστολής της πληρωμής. Οπότε έχουμε αμέσως ροή πληρωμής. Ε, αν δηλαδή έχουμε πάρει κάποιες, ε, ε, έχουμε κάποιες αξιώσεις για πληρωμές στον τομέα αυτό που σας είπα, τον μεταφορών και έχουμε πληρώσει το 5% για παράδειγμα. Τότε μπορούμε, επειδή αυτές οι δαπάνες πρέπει να καταβληθούν, μπορούμε τότε να δώσουμε αυτά τα κονδύλια και άμεσα. On Επί του θέματος που ετέθη από την Αυστριακή συνάδελφο σε σχέση με την εταιρική σχέση. Και αυτό συνδέεται με αυτό που είπε ο κύριος Ζήλα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το θέμα του ξαναεπαναπρογραμματισμού απαιτεί μία συμφωνία της ε, Επιτροπής Εποπτείας για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει η Επιτροπή η οποία εποπτεύει το σχέδιο αυτό να εγκρίνει την ε, απόφαση αλλαγής του λειτουργικού σχεδίου, του λειτουργικού προγράμματος. Και μέσα σε αυτή την ε, ε Επιτροπή Παρακολούθησης έχετε όλους τους εμπλεκομένους κυρία Ζέλα τώρα για τις ε, διασφαλίσεις προς όφελος των περιφερειών. Ιδίως όταν πρόκειται για το θέμα ορισμένων σχεδιών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ατενίσει κανείς με προσοχή όταν εφαρμόζει αυτήν την ε, αίτηση για τον ε, παραπρογραμματισμό μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη λοιπόν πρόταση. Μπορεί κάποιος να θέλει απλώς να εξασφαλίσει, να θέλει εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση αυτών τα οποία είναι υπό εφαρμογή. Από ό,τι κατανοώ όμως, <clears throat> αυτό το θέμα θα πρέπει να διαλευκανθεί μέσω του διαλόγου, ο οποίος προβλέπεται μεταξύ Κομισιών και Κρατών Μελών και όλος ιδιαίτερος η απάντηση του κράτους μέλους σε μια τέτοια έκκληση προγραμματισμού θα πρέπει να εξηγεί πώς θα ληφθούν υπόψη οι διασφαλίσεις για τις περιφέρειες και πώς θα αντιμετωπιστεί ο, αντι, ο αντικός δυνητικά αντίκτυπος ο οποίος θα μπορούσε να αποκλειθεί. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτό. Και επίσης ό,τι πρόκειται για τις εθνικές προτεραιότητες και κατά πόσον οι εθνικές προτεραιότητες μπορούν να παίξουν και κάποιο ρόλο στην αλλαγή προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να κρατάτε στο μυαλό σας το γεγονός ότι η επιλογή αυτή επαναπρογραμματισμού έχει νόημα μόνο όταν έχει να κάνει με κινητοποίηση χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα για ένα κράτος μέλος το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο έχει διαφανεί από μια ε, σύσταση ειδική για τη χώρα αυτή, ένα κάτω μέλο μπορεί πάντα να κινητοποιήσει άλλε μορφές υποστήριξης. Αν λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συστάσεις αυτές με καθαρά εθνικά μέτρα, αυτό δεν καθιστά απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία του άρθρου 23 και να έχουμε μια αίτηση που αφορά τον προγραμματισμό και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας και τις απαντήσεις σας. Ας δούμε τι θα γίνει με τις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα για να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες από την Κομισιόν. Μπορούμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την μέλησια διάταξή μας. Τώρα έχουμε την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Οι συντονιστές συναντήθηκαν χθες το βράδυ και οι αποφάσεις τους απεστάλησαν σε εσά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρέπει να τις εγκρίνουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Σας ευχαριστώ για αυτό. Εγκρίνουμε λοιπόν τις αποφάσεις των συντονιστών. Το επόμενο σημείο είναι τα διάφορα. Έχουμε διάφορα. Όχι, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε χωρίς τα διάφορα. Και το τελευταίο σημείο είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Πρέπει να σας πληροφορήσω ότι η επόμενη συνεδρίαση προβλεπόταν για τη Δευτέρα και την Τρίτη 6 και 7 Οκτωβρίου. Αλλά ένεκα της ακρόασης του Αντιπροέδρου κυρίου Τίμερμανς που θα λάβει η χώρα το πρωί της 7ης, της 7ης μάλλον Οκτωβρίου με το σχήμα ανοιχτή συνεδρίασης των Προέδρων των πολιτικών ομάδων ως λέγουν οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να υπάρχουν παράλληλες συνεδριάσεις επομένως θα πρέπει να ακυρώσουμε τη συνεδρίασή μας για το πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Η συνεδρίασή μας της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, το απόγευμα της 6 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί όμως και έχουμε μια ειδική ημερήσια διάταξη για αυτή την συνάντηση, η οποία θα αφιερωθεί σε μια κοινή ε, συνάντηση με την ομόλογη μας επιτροπή στην Επιτροπή των Περιφερειών. Θα είναι το πρώτο τμήμα της Ευρωπαϊκής, η πρώτη μέρα μάλλον της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Πόλεων που είναι ένα γεγονός το οποίο συνδιοργανώνεται από την Κομισιόν και την Επιτροπή των Περιφερειών. Λεπτομεριακό πρόγραμμα για τη συνάντηση της 6 Οκτωβρίου θα αποσταλεί αργοτέρως. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την εργασία τους και την εγκαρτέρησή τους χθες και σήμερα και κλείνω τη συνεδρία της Επιτροπής μας.